και κύριοι σας καλοχαιρετίζω. Liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλοχαιρετίζω. Ζήτω πρώτα συγγνώμη που καθυστέρησα να φτάσω. Μου συμβαίνει σχετικά σπάνια, όπως γνωρίζετε, να καθυστερώ. Αλλά είχα υποσχεθεί σε αυτή τη διάσκεψη των δημάρχων να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Και η ο προλαλής σας από ένα πεντάλεπτο παρέμβασης έκανε μια παρουσίαση δηλώσεων επί των αρχών. Και είχα δυσκολία, δεν μπορούσα να φύγω, έπρεπε να παραμείνω καθυστέρησα. Ζητώ συγγνώμη. Περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Αν θέλετε που αναβάλαμε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για το ψήφισμα μπορούμε σχετικά σύντομα να ολοκληρώσουμε. Απλά να ψηφίσουμε χρειάζεται αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Λοιπόν, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Εντάξει, συμφωνείτε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Δεν έχετε κάρτα εσείς. Εντάξει, ένας. θα προσμετρήσουμε την ψήφο σας μετά εκ των υστέρων. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Εκείνοι που... Ε, δεν θα αρχίσουμε διαδικαστικά. Κλωτούρμες. Sure. Ε, Για να με βέβαιος τι κάνουμε. Εκείνοι που είναι με τον Παρ των τον Σβόμποντα και με μένα που είμαστε υπέρ του ψηφίσματος. Αυτό θα κάνουμε τώρα, έτσι. Θα δούμε αν είμαστε υπέρ ή κατά. Λοιπόν, είναι σχετικά απλό. Όσοι είναι υπέρ του ψηφίσματος θα ψηφίσουν με ναι. Θα υπερψηφίσουν. Όσοι είναι κατά θα καταψηφίσουν με όχι. Είναι στην φύση των πραγμάτων. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι και απλό κιόλα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και τους άλλους συναδέλφους θα τους καταμετρήσω αργότερα. Συμφωνείτε? Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Δεν υπάρχουν παραπάνω ψήφοι πέρας ψηφοφορίας διαμαρτυρία. Closed. Πέρας ψηφοφορίας, εντάξει. Όχι, με τους Ολλανδούς τι γίνεται. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε, ακυρώνουμε την προηγούμενη ψηφοφορία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το ξανακάνουμε, θα επαναλάβουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι λοιπόν. E ένας από το ΕΛΚ παραπάνω, ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα, πέρας ψηφοφορία, συμφωνείτε. Ωραία. Πλειοψηφικά απορρίφθηκε τώρα. Τώρα όμως θα προσμετρήσουμε τις ψήφους εκείνων ποιοι ήταν υπέρ και... Λοιπόν, 20 υπέρ. 20 υπέρ. Μαντουρέλ εσείς, κυρία Μαντουρέλ. Α, εντάξει, ωραία. 20 υπέρ 23 εναντίον λοιπόν. Και έτσι απορρίφθηκε το ψήφισμα. Τελείωσε και πάει και ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και φιλικότητα και ικανοποίηση και όλα τα άλλα τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ενέργειας Τις τελευταίες ημέρες αυτό που είχαμε πει ήταν μετά την εκλογή τώρα του Επιτρόπου θα συζητούσαμε για το σχέδιο εργασίας του και το, το πρόγραμμά του. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Χωρίς τώρα μεγάλες εισαγωγές και εισαγωγικούς λόγους θα περάσουμε στην ουσία. Θα μου ευγνώμων αν υπήρχε κάποια ησυχία στην αίθουσα για να ξεκινήσει ο Επίτροπος. Κύριε Επίτροπο, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για το ότι μου δίνετε την πρώτη ευκαιρία αυτή να είμαι παρόν σε σχέση με την ακρόαση μαζί σας να περνάμε τώρα σε μια συζήτηση. Τις τελευταίες εβδομάδες είχα κάποια διμερεί θέματα που συζήτησα μαζί σας και με τους επιμέρους ε, εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων Είχα σημαντικές προτάσεις, αξιόλογες προτάσεις που υποβάλατε και εκείνους τους βουλευτές που δεν μπόρεσα να συζητήσω μαζί τους, τους προσφέρω όποτε επιθυμούν κατηδίαν να μπορέσουμε να συζητήσουμε άτυπα κάποια θέματα. Είναι σημαντικό αυτό νομίζω. Σημαντικό για να έχουμε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή εταιρική σχέση και να υπάρχει πληροφόρηση για το τι κάνουμε σε σχέση με το έργο μας σε αυτές τις άτυπες συζητήσεις. Και τώρα είμαι στη διάθεση όλων φυσικά και προσκαλώ όλους σας να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Όλη η Επιτροπή, το σύνολο της Επιτροπής, τα θέματα τα ενεργειακά τα, έχει, έχουμε εγγράψει πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Αυτό δείχνει και η δράση των κρατών, οι δηλώσεις και δεσμεύσει του Προέδρου συζητήσεις της Επιτροπής μας με άλλες κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο πρόσφατα, όπου η προστασία του κλίματος και τα ενεργειακά θέματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους Κινέζους που έδειξαν ενδιαφέρον και προθυμία να συνεχίσουν την εταιρική σχέση μαζί μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για κατεπήγοντα θέματα όπως τον Αμπούκο, τον πετρελαγωγό, αεραγωγό σαφή μηνύματα να προχωρήσουμε με τη δημιουργία ηλεκτρικών οχημάτων και προετοιμαζόμαστε τώρα <clears throat> για τα κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με κάποιο καλό τρόπο ώστε αποκινούμε το Κοινοβούλιο να βρούμε νέες χρήσεις κατά τη διάρκεια <clears throat> του έτους μέχρι τα τέλη του έτους. Μακροπρόθεσμες δραστηριότητες είναι η στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως φυσικά και το πρόγραμμα δράσης για τα θέματα ενέργειας, θα επανέλθω σε αυτό, και οι οδικοί χάρτες ε, για το 2050. Σας προσκαλώ γι' αυτό, Ρίτα, να διαβουλευτούμε από κοινού και να καθορίσετε τις θέσεις σας για τη, για, το, για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική και τον προγραμματισμό της για όλους τους εμπλεκόμενους για τις επόμενες δεκαετίες ε, η συμμετοχή όλων είναι πολύ σημαντική. Κύρια στοιχεία θα είναι η διαδικτύωση στα δίκτυα υποδομών, τεχνολογία στη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και διοξιδίου του άνθρακα και επίσης ε, η πολυμορφοποίηση ενεργειακών πηγών και πόρων και υποδομών έναντι της σημερινής κατάστασης και εξάρτησης στην οποία βρισκόμαστε. Επιτρέψτε μου σύντομα σημαντικά έργα να σκιαγραφίσω που αφορούν ε, το κοινό μας έργο που θέλουμε από κοινού να επιτελέσουμε. Πρώτα απ' όλα η πλήρης ε, ε, τροποποίηση και αλλαγή της νομοθεσίας στην ενιαία εσωτερική αγορά. Περαιτέρω νομοθετικό έργο. <clears throat> Εκτέλεση και εφαρμογή ενισχύει διατάξεων στην πρακτική εφαρμογή. Η ενιαία εσωτερική αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο βρίσκεται στη σωστή πορεία, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά έναντι στα όσα έχουν γίνει με άλλα αγαθά και εμπορεύματα <clears throat> και δεν έχουμε σημειώσει επαρκή πρόοδο για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον, δημιουργία σταθερών συνθήκων πλαισίου και πολυμορφοποίηση για τις υποδομές των δικτύων και των δικτύων υποδομών τα δίκτυα υποδομή για τα αέρια με την αλληλεγγύη, αυτό είναι σημαντική έννοια, και μείωση της εξάρτηση. Επίσης ε, για την ηλεκτρική ενέργεια θα είναι κέριο βάρο κεντρικό σημείο ε, των εργασιών μας. Το λέω και πάλι, χωρίς να δεσμεύομαι με λεπτομέρειες, εσείς θα πρέπει από κοινού μαζί μα να συναποφασίσατε αν μετά το έκτακτο πρόγραμμα που γεννήθηκε μέσα στην κρίση των οικονομιών μας, θα έχουμε μια αηφορία και συνέχεια αηφόρο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος με τη διεύρυνση των υποδομών μας για τα ενεργειακά θέματα και αν και πώς θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μεταξύ των κρατών μελών και προς τα κράτη-μέλη και ολοκλήρωση και ε, ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις υποδομές για την μεταφορά αυτών των ενεργειακών ε, προϊόντων από την πηγή μέχρι τους καταναλωτές. Offshore αιωλικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα. Υποδομή και δίκτυο ευρωπαϊκό που θα συνδεθεί με αυτές τις πηγές. Χωρίς υποδομές και δίκτυο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Για την υποδομή υπάρχει σαφής σειρά και απαρίθμηση πραγμάτων. Πρώτον, οι ιδιοκτήτες, οι κύριοι που θα έχουν την κυριότητα των δικτύων, επιχειρήσεις ενεργειακές και άλλες. Έτσι, δεύτερον, θα έχουμε τις, αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές που θα μπορέσουν να ασκήσουν κέριο ρυθμιστικό ρόλο και σε περαιτέρω α, λειτουργία της δικής μας ρυθμιστικής αρχής που θα, αρχίσει να, θα συνεχίσει το έργο της και που με αυτή τη στιγμή πρέπει να επιλέξουμε το Γενικό Διευθυντή της, θα έχουμε αποφασιστικό ρόλο που θα διαδραματίσει ρόλο ολοκλήρωσης και αφομοίωσης. Ξεκινάμε με μεγάλες προσδοκίες. Δεν αποκλείουμε η ΕΣΑ κατά τη διάρκεια των επομένων ετών να ενισχυθεί όσον αφορά τις αρμοδιότητές της και να χρειαστεί ενίσχυση αρμοδιοτήτων. Όσον αφορά τον ενιαίο εναέριο χώρο που γίνεται δεκτός ως ανάγκη σήμερα, αυτό θα μπορούσε να είναι γνώμονας ώστε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο διασυνοριακά. Και τρίτον, επίσης, πιστεύω ότι μια συμπληρωματική δράση όσον αφορά την συγχρηματοδότηση με κίνητρα που θα δίνουμε εκεί όπου οι ποδομέσα δεν είναι κερδοφόρες στα δίκτυα, όμως χρειάζονται κατεπηγόντως οι υποδομές των δικτύων εκεί με κίνητρα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα συνέχισης του προγραμμάτός μας ε, τις επόμενες δεκαετίες και αξίζει να προβληματιστούμε να δούμε τι θα κάνουμε μακροπρόθεσμα. Προσφέρουμε στην Ευρωβουλή αυτή την εμπλοκή και συναπόφαση μαζί μας για αυτά τα θέματα. Μετά θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο την πρόθεση των στόχων της στρατηγικής 2020 στις εκπομπές ρήπων και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να θέσουμε κέντρο βάρους στα, στη βιομηχανία και ε, στην έρευνα. Πανευρωπαϊκές προσπάθειες για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και επιδόσεων, επίσης ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας και οι βέλτιστες ανώτατες προδιαγραφές για την ε, ατομική ενέργεια. Επίσης, αυστηρές προδιαγραφές για τα απόβλητα, τα πυρηνικά απόβλητα. Προετοιμάζουμε ένα σχέδιο για νομική ρύθμιση για την τελική αποθήκευση των ραδιενεργών αυτών αποβλήτων. Και έτσι από κοινού μαζί σας το φθινόπωρο θα ξεκινήσουμε διάλογο μαζί σας για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται επίσης και για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρικής σχέσης με τις χώρες που παράγουν και εξάγουν ε, ενεργειακούς πόρους και προϊόντα. Πρέπει να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία. Το Ναμπούκο, ο Ναβουχοδονόσορας είναι ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης στους βουλευτές, στους ευρωβουλευτές από τα κράτη-μέλη να στραφώ, από τα οποία κράτη θα περάσει αυτός ο αγωγός βλέπω με σεβασμό πως κάποιοι εμπλεκόμενοι <clears throat> ε, stakeholder είναι υπέρ του South Stream. Θέλω να παρακαλέσω όλα τα κράτη-μέλη στην προοπτική του Ναμπούκο να παραμείνουμε πιστοί εφέτος. <clears throat> Διότι όταν έχουμε μεγαλύτερες υποδομές υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό ισχύει για το North Stream, αλλά μόνο το Ναμπούκο μας φέρνει πιο κοντά σε σχέση με το, τη διάθεση φυσικού αερίου και γι' αυτό αυξάνεται η ασφάλειά μας, μειώνεται η εξάρτησή μας. Μόνο όταν όλα τα κράτη-μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι, ευρωβουλευτές θα είναι αλόβητοι και δεν θα, μπορούν, δεν θα ε, καμφθούν, μόνο τότε το Ναμπούκο θα μπορέσει εφέτος να καταλήξει σε απόφαση και απόφαση για την εκτέλεση των ε, έργων του. Η ενεργειακή μας πολιτική είναι ακριβώς η προσπάθεια για την ευρωπαϊκή οικονομία και την αηφορία και ασφάλεια των καταναλωτών να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές τρύπων. Αυτό πρέπει να είναι η κοινή μας δέσμευση και αυτή πρέπει να προάγουμε. Για να καταφέρουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε μια ενιαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική που θα βασίζεται σε ένα νέο πρόγραμμα δράσης από πλευράς μας. Το νέο ενεργειακό πρόγραμμα δράσης έχει και τον οδικό χάρτη για το 2050 για την μείωση των εκπομπών ρήπων από τον άνθρακα, μείωση της χρήσης του άνθρακα. Συνειδητά τώρα δεν πρέπει να επιλέξουμε μια βιαστική και λίγο όρημη και ανώριμη πολιτική αλλά πρέπει με σύνεση και σοφροσύνη να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας γι' αυτό. Το νέο πρόγραμμα δράσης ε, θα είναι ένα πρακτικό μεσοπρόθεσμο μέσο ή εργαλείο που θα μας δίνει τη δυνατότητα τους στόχους του 2020 στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική να τους πετύχουμε. Θέτει προτεραιότητες ε, και θα έχουμε στην πρόοδο της εξέλιξης των έργων την ε, εποπτεία, την επιτήρησή τους. Θα έχουμε ένα ευρύτατο πλαίσιο πολιτικών στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διασφαλίζουμε έτσι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το μικρότερο κόστος και το μεγαλύτερο κέρδος, το μέγιστο κέρδος θα μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πολιτική που πρέπει να την ακολουθήσει με επιτυχία. Η στρατηγική στα κράτη-μέλη και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο θα επεκτείνεται, ώστε να μπορεί να διασφαλίσεται η αηφορία πανευρωπαϊκά και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στην ε, διάσκεψη των δημάρχων που γίνεται εδώ ταυτόχρονα και θα εξακολουθήσει τις επόμενες δύο θα διαρκέσει δύο ημέρες. Έχουμε τους τοπικούς εκπροσώπους ε, δήμων και κοινοτήτων, δημάρχους. Είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει ότι η Ευρώπη παντού μπορεί και ασχολείται και πρέπει να ασχολείται με αυτά τα θέματα ώστε να προαθούν όπως πρέπει. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους θέλω σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες να ζητήσω να συνεισφέρουν από πλευράς τους. Γι' αυτό θα έχουμε ένα έγγραφο συζήτησης, μια επισκόπηση ε, των πραγμάτων ως έχουν σήμερα και αυτό θα προπαρασκευάζει τα σχετικά με το πρόγραμμα ενέργειας που έχουμε, το ενεργειακό μας πρόγραμμα και θα είναι και η βάση για τη συζήτηση των Υπουργών Ενέργειας ε, που θα διεξαχθεί τον Μάιο. Η εικόνα της κατάστασης αυτή που θα υποβληθεί θα είναι μια κριτική αξιολόγηση όλων εκείνων που από την έγκριση του πρώτου ενεργειακού προγράμματος δράσης πετύχαμε, αλλά και αυτών που δεν πετύχαμε ακόμα. Δεύτερον, θα δείξει ποια είναι τα κενά και τα χάσματα που υπάρχουν, όπου περαιτέρω μέτρα απαιτούνται να ληφθούν σε σχέση με την, με οικονομία, ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, νέων πρωτοβουλειών με νέες βάσεις. Περισσότερες προτεραιότητες θα παριθμούνται που θα μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων μας. Θα καλύπτει την ανάγκη, την αναγκαιότητα πλήρους εφαρμογής των μέτρων αυτών και θα τονίζει την λήψη αυτών των μέτρων. Η ασφάλεια ανεφοδιασμού σε ενεργειακά προϊόντα, η αηφορία, η επίτευξη της στρατηγικής 2020 είναι απαραίτητα στοιχεία που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και η χρηματοδότηση είναι ένα θεμελιώδες θέμα για τα ενεργειακά ζητήματα. Υποχρηματοδότηση εννοώ αφενός ενέργεια, έρευνα, δεύτερον ενεργειακά προγράμματα με τους εταίρους μας, τρίτον συγχρηματοδότηση. Χρηματοδότηση όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα υποδομών. Να μην αυταπατώμαστε. Έτσι ξεκινά μια συζήτηση επί των θεμελίων για την επόμενη περίοδο και για το ποιο ρόλο θα διαδραματίζει η ενέργεια, τα ενεργειακά θέματα μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Θέλω να ακούσω, αδειμονώ να ακούσω και να σημειώσω τις απόψεις σας. Το έγγραφο θα τύχει ευρεία ε, δημόσια διαβούλευση ε, και θα δώσει κίνητρα για να προαχθεί αυτό ο διάλογο. Και έτσι είσαστε εσεί ο πρώτο εταίρο στι διαβουλεύσεις αυτέ για μας. Το ενεργειακό πρόγραμμα δράση, σύμφωνα με το σχεδιασμό μα, θα ε, εγκριθεί τελεσίδικα τον Ιανουάριο. Έχουμε περίπου ένα εξάμεινο το οποίο θα αφιερώσουμε σε διαβουλεύσεις μέχρι να οριμάσουν τα πράγματα και να εγκριθεί τελεσίδικα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2011 θα υποβληθούν περαιτέρω μέτρα. Θέλουμε να προτείνουμε ένα ονοδικό χάρτη που τα διαφορετικά σενάρια για την αηφορία θα τα εξετάζει. Για μια σε χαμηλή χρήση άνθρακα οικονομίας μέχρι το 2050 θα προβλέπει με τα ορόσημα και τα, τις αναγκαίες δράσεις. Να περάσουμε σε ένα νέο σύστημα, σε μια κοινή προσέγγιση, μακροπρόθεσμα, με στόχους και μέσα που θα καθοριστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι. Μέσα σε αυτό ανήκει η προσπάθεια, η, την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα να την μειώσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πόρων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας. Πρέπει στόχος να είναι η αηφορία και να έχουμε έτσι την βέλτιστη χρήση με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας <clears throat> με την αποθήκευση που θα διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο και όπου θα είναι αναγκαίο και όπου εθνικά θα επιθυμείτε αυτό <clears throat> μπορεί να υπάρξει ένα μείγμα ενεργειακών πηγών με την χρήση και ατομικής ενέργειας που σήμερα <clears throat> περίπου παράγει η πυρηνική ενέργεια τα δύο τρίτα της χαμηλής εκπομπές ρήπων τεχνολογία, με τη χαμηλής εκπομπές ρήπων τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένων των ε, ε, θεμάτων υποδομής ε, και των, της των στενοπών που παρακολύουν την καλή λειτουργία τη της ενιαίας ενεργειακής αγοράς θα προτείνουμε ένα ενεργειακό πρόγραμμα υποδομών με βάση τα, την πείρα μας και την πολιτική μας με το GNPR. Θα καθορίσουμε προτεραιότητες για τις υποδομές, για τα ενεργειακά δίκτυα για τις επόμενες δεκαετίες. Και τέλος προς το συμφέρον <clears throat> σαφών προοπτικών για την καινοτομία το πακέτο για την ανακοίνωση αυτή θα προβλέπει προτεραιότητες για τις επόμενες δεκαετίες και μια ανακοίνωση για τις ρυθμιστικές δράσεις και τα μέσα που θα χρειαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Για τις 28 Μαΐου έχουμε προβλέψει με την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου μια διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη και όπου <clears throat> και τους ευρωβουλευτές προσκαλούμε να συμμετάσχουν πριν από τα τέλη του 2010 το πακέτο αυτό θα έχει εγκριθεί. Αυτό είναι ο στόχος μας. Η πείρα με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομικής συγκυρίας μέχρι σήμερα πήγε πολύ καλά, πολύ ικανοποιητικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον ε, προηγούμενο επίτροπο και σήμερα που έχω αναλάβει εγώ τη σκητάλη ήταν σε θέση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο να διασφαλίσει κινητοποίηση πολλών μεγάλων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση. Και μέσω αυτών των δράσεων έχουμε ξεκινήσει για τις υποδομές ε, τα αναγκαία μέτρα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια τροποποιητική πρόταση που θα υποβάλουμε που την ανακατανομή των μη καταβληθέντων, μη δαπανηθέντων κονδυλίων <clears throat> μέσα στο πλαίσιο αυτών των δράσεων θα, προβλέπουν, θα προβλέπετε πώς θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη χρήση της ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη για μια ταχεία έγκριση αυτής της πρότασης, ώστε η διαδικασία αυτή μέχρι τα τέλη του έτους να μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί και έτσι να αποφύγουμε μια διαγραφή κονδυλίων, μια διαγραφή της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης κονδυλίων. Εδώ η προϋπόθεση είναι επιθυμητή να υπάρξει εμπλοκή και του τοπικού επίπεδου και περιφερειακού επίπεδου. Έτσι με ένα ευρώ παράγουμε υπεραξία επιτόπου στους δήμους, στις κοινότητες, επιτόπου στις περιφέρειες. Αυτό με φέρνει και με οδηγεί σε ένα άλλο περαιτέρω συγκεκριμένο βήμα η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένας τομέας που και για σας ευρωβουλευτές και για μένα είναι πολύ σημαντικός. Γι' αυτό εργαζόμαστε σε, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την βέλτιστη αποδοτικότητα της χρήσης των ενεργειακών πόρων με τα αναγκαία μέτρα που θα προβλέπονται. Κύριοι στόχοι αυτής της στρατηγικής για την αποδοτικότητα της ενέργειας είναι η αποδοτικότητα να είναι ένα κύριο τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών και έτσι να κατοχυρώνεται και να είναι μέρος των άλλων συναρμόδιων και συναφών πολιτικών επιλογών. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την αποδοτικότητα των ενεργειακών πόρων θα πρέπει μέχρι τα τέλη αυτού του έτους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο αρχές 2011 με ένα τεχνικό έγγραφο που θα συμπληρώνει αυτές τις πτυχές να εγκριθεί. Η αξιολόγηση αυτή είναι μέρος ενός πακέτου που ακριβώς ε, για τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ε, μέχρι το 2020 αυτής της στρατηγικής θα διαμορφώνει πλαίσια για την επίτευξη των στόχων. Αυτά τα ορόσημα και ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής μας θέλω να αναφέρω. Μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε πρόταση για την αντιμετώπιση των πυρηνικών αποβλήτων και των καμένων ράβδων από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και έτσι με υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οδηγία αυτή για την πυρηνική ασφάλεια που επετεύχθη ήταν ένα βήμα ώστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ομοιογενές πλαίσιο για την πρόθεση των προϋποθέσεων αυτών. Αν ασχοληθούμε μόνο για απόβλητα από τα, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες από την έρευνα και από την ιατρική θα είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος ώστε από πλευράς της Ευρωβουλής αυτή η νέα προώθηση να ακολουθηθεί. Εδώ δεν πρόκειται μόνο και θέλω να το τονίσω αυτό για το θεμελιώδες θέμα υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είναι απόφαση των κρατών μελών, των εθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων. Εδώ όμως πρόκειται για την κοινή μας ευθύνη για την ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την τελική αποθήκευση αυτών των πυρηνικών αποβλήτων. Θέλω να προσθέσω εδώ, για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε σωστά το έργο μας, τα καθήκοντά μας και να μην ασχολούμαστε με εξαγωγές και άλλους πειρασμούς που μπορεί να είναι θελκτικοί και να επιλέγουμε πού θα αποθηκεύσουμε αυτά τα προϊόντα κάπου στο εξωτερικό. Επίσης με αυτή την πρόταση όπως και ε, ο κανονισμός για την ασφάλεια ε, επάρκειας ε, με το φυσικό αέριο και την ενεργειακή διασφάλιση όλα αυτά τα βήματα θα οδηγήσουν την ενεργειακή μας πολιτική ένα βήμα παραπέρα και ενδιαφέρομαι σε στενή συνεργασία μαζί σας να γίνουν αυτά όχι βιαστικά αλλά αντικειμενικά νυφάλια, ήρεμα και είμαι βέβαιος, τέλος πρέπει να πω, ότι με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία ευρωπαϊσμού, εξευρωπαϊσμού των ενεργειακών πολιτικών θα είναι σε καλή οδό, σε καλή πορεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε Έτσιγκα για την διεξοδική περιεκτική αυτή παρουσίαση των εργασιών των επόμενων μηνών από την Επιτροπή. Τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα εδώ δεν θα συζητήσουμε σε βάθος και σε εύρος όλα τα σημεία. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι δυνατόν. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι ότι 18 έχουν ζητήσει τον λόγο να παρέμβουν. Αυτό υποχρεωτικά με οδηγεί στο αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να πρέπει να πούμε ότι ευθύ εξ αρχή θα συμφωνήσουμε καθένας θα προσπαθήσει με ένα λεπτό να πει αυτά που έχει να πει. Γιατί διαφορετικά κάποιοι συνάδελφοι μετά δεν θα έχουν χρόνο να διατυπώσουν ερωτήσεις. Μας ενδιαφέρουν και οι απαντήσεις έτσι από τον Επίτροπο. Και για αυτά τα 18 ερωτήματα χρειαζόμαστε κάποια λίγα λεπτά να απαντήσει ο Επίτροπος. Θα ήμουν ευγνώμων να προσπαθήσετε σε ένα λεπτό να καλύψετε τις ανάγκες σας. Με κάθε ευγένεια. Να τα, ό,τι είναι περιττό να μην το αναφέρετε ευγένειες, φιλοφροσύνες, στο θέμα και στην ουσία να επικεντρωθείτε και όχι σε φιλοφροσύνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Ως πρώτος η κυρία Κολόσκα, Κολόσκα Βίσκα έχει τον λόγο. Πού είναι, εκεί. Παρακαλώ εσείς, είσαστε οι πρώτοι. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε φιλοφρονήσεις, ε, στο συγγνώμη. Περνάω στην ουσία. Κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας απαντήσατε σε μία από την ερώτησή μου όσον αφορά το North Stream, ότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή ελληνική για τη συμφωνία αυτή και υποσχεθήκατε τότε ότι θα εφαρμόσετε την ευρωπαϊκή ελληνική σύμφωνα με τα άρθρα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είπατε επίσης ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τις διμερείς συμφωνίες και να περάσουμε σε ευρωπαϊκές συμφωνίες. Παράλληλα, συμμετείχατε στην επίσημη έναρξη του αγωγού Nord Stream. Κύριε Επίτροπε, έχω την εξής ερώτηση. Θα ήσασταν υπέρ μιας Ευρωπαϊκής κυβερνητικής Συμφωνίας πέρα από τις εμπορικές συμφωνίες όσον αφορά το Nord Stream, όπως ακριβώς υπάρχει και στην περίπτωση του Ναμπούκο. Επίσης, θα το προσθέτατε αυτό ουσιαστικά στο πρόγραμμά σας για τα επόμενα χρόνια ώστε να υπάρχει μια διαφανής τέτοια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να κάνει το Nord Stream ένα πραγματικά ευρωπαϊκό φυσικό αγωγό, αγωγό φυσικού αερίου και κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγαμε κάποιες από τις ρήτες που υπάρχουν στην τρέχουσα συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κρίστιαν Έλερ τώρα παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, χωρίς φιλοφροσύνες τώρα άμεσα στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε δημοσιεύματα όπου τονίζω καταρχήν έλεγαν και ανέφεραν ότι για τους αντιδραστήρες, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας δεν πιστεύετε σε αυτά που στη Γερμανία ή ευρωπαϊκά θα έχουν χαμηλές εκπομπές ρήπων. Τώρα τι γίνεται με τις πιλωτικές αυτές εγκαταστάσεις ε, δισεκατομμυρίων. Η τοποθέτησή σας ε, για τους συναδέλφους ε, που είχαν αυτές τις θέσεις δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας σε σχέση με αυτό το ζήτημα δεδομένου του ότι για την έκθεση Stern αναφέρθηκε ότι με την τεχνολογία αυτή δεν θα μπορέσει να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων του 2020. Κλωτούρμες παρακαλώ. Κλωτούρμες, bist έχετε τον λόγο. Εσύ έχεις τον λόγο, Κλοντ. Άλλη έκπληξη. Θα ήθελα να συγχαρώ για τα 115 εκατομμύρια για κάθε ευρώ από αυτά για τις πόλεις, δήμους και κοινότητες. Μία ερώτηση τώρα για τα καλώδια και αν διαπιστωνόταν ότι στην άλλη πλευρά της Μεσογείου για το Desert Tech ε, θα είχαμε ε, με παράκαμψη του ETS παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα λέγατε ότι αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεύτερον Ευρωπαϊκή ε, ο Οδικός Χάρτης για το 2020 άκουσα ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η δική σας υπάλληλη δηλαδή, εργάζονται και υπολογίζουν ένα σενάριο με 75% μείωσης ε, διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Μας εξέπληξε αυτό, διότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν πει 80 ή 90% αυτή η μείωση, αν θέλουμε να πετύχουμε την μείωση της αναθέρμανσης του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα τι γίνεται με τους οδικούς χάρτες. Ακούσαμε ότι σε σχέση με κάποια σενάρια ε, διακύμανσης από τον καθηγητή Χάτφους είχαν γίνει αυτά. Και ο ίδιος είχε παρουσιάσει ένα αμφίσιμο σενάριο, ε, αμφιλεγόμενο σενάριο όπου υποχρε... πολύ, πολύ γοργά, ας το πω έτσι, ε, προβλεπόντουσαν κάποια μέτρα. Και εντάχει το Γαλλικό Κοινοβούλιο σήμερα θα αποφασίσει κάτι εξαιρετικό και αν αποφασίσουν ότι για τις εολικές ενέργειες, ε, για την αιωλική ενέργεια στη Γαλλία θα πρέπει να υπάρχει και κατάθεση ε, εγγυητικών επιστολών στις τράπεζες. Δεν θα ήταν μια τέτοια καλή ιδέα να γίνεται το ίδιο και με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η κυρία Τικάου παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαι κυρία Επιτροπέ. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Οπωσδήποτε ήθελα να τονίσω και εγώ την σημασία του προγράμματος Ναμπούκο. Είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ούτε περιθώριο για ερωτηματικά εδώ. Όμως εγώ ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που κι εσείς στην παρουσίασή σας. Δηλαδή, ότι θα υπάρξουν πόροι από τα διευθυντικά, από τα ταμεία μάλλον της οικονομικής αναδιάρθρωσης, τα οποία δεν θα έχουν αξιοποιηθεί, πόροι που δεν θα έχουν αξιοποιηθεί και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν. Ξέρουμε ότι στον κανονισμό αυτού του ταμείου υπάρχει η πρωτοβουλία Smart Cities, μεταξύ άλλων. Ελπίζω λοιπόν, μεταξύ των μεριμνών σας, να βρεθεί και αυτή, οι επενδύσεις δηλαδή, για να βελτιωθεί ενεργητική, η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Ελπίζω ότι αυτή η προτεραιότητα θα σας απασχολήσει στο μέλλον και ότι θα αυξηθούν οι πόροι προς αυτό το σκοπό. Σε ευχαριστώ. Συνάδελφος Έντσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην σας συγχαρώ για το έργο σας από τη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, από την ακρόασή σας δηλαδή ως σήμερα. Και αυτό γιατί πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που κατά την ακρόαση είχαν και κάποιους ενδιασμούς. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Και δεδομένου ότι όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν το ίδιο δυναμικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγου χάρη, για την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια και ούτω καθεξής, και δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ήθελα ο Επίτροπος αν μπορεί να μου απαντήσει στο εξή. Έχει σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα στήριξης των 100 μελών για να οικοδομήσουν και να ανανεώσουν τις υδροηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις Αυτέ που υπάρχουν σε ορισμένε χώρες ή ενδεχομένω να οικοδομήσουν νέες τέτοιες εγκαταστάσεις, εργοστάσια υδροελεκτρική ενέργειας και προκειμένου να δώσουν τέρμα στη χρήση των εργοστασίων που κινούνται με τον άνθρακα. Σα ευχαριστώ κυρία Καρβάλιο, παρακαλώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, παρόλο το γεγονός ότι τα ενεργειακά θέματα έχουν πολιτική προτεραιότητα σήμερα, τα κονδύλια για την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας και επίδειξης όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι πιο περιορισμένα από ότι για παράδειγμα στην δεκαετία του 80. Τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση για την προπαρασκευή του 8ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη και επίδειξη και θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το πρόγραμμά σας, για την έρευνα, για τα ενεργειακά θέματα και πώς θα χρηματοδοτηθούν και ποιες προτεραιότητες. Θα βασίζονται οι προτεραιότητες στις λύσεις και απαντήσεις των μεγάλων προκλήσεων και θα βασίζονται σε τεχνολογικές προοπτικές και ποιες θα ήθελα να μας σχολιάσετε τι θα γίνει με την τεχνολογία των προγραμμάτων και εγχειρημάτων επίδειξης, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ποια θα είναι τα προγράμματα επίδειξης και πιλωτικά προγράμματα στο νέο αυτό πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ο Κυρία Herzog, παρακαλώ. Yes, ε, Thanks, ε, thanks very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου για μια πολύ σύντομη ερώτηση. Πρώτον, εξ ονόματος Επιτροπής μας, ενδιαφερόμαστε για το πώς θα ασκήσετε πίεση προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί περισσότερο η υπηρεσία ΙΣΕΡ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις μέχρι το 2050 σε προγράμματα οικονομίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο όμως περιβάλλον προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αυτές επενδύσεις. Τρίτον, όσον αφορά την έρευνα. Θα προωθήσετε και άλλα προγράμματα ερευνητικά σαν αυτά τα οποία αναφέρατε ή θα επικεντρωθείτε περισσότερο στο ΙΤΕΡ και τι μορφή θα πάρουν τα προγράμματα ΙΤΕΡ. Πήγατε στο Αζερβαϊτζάν, εκτιμήθηκε ιδιαίτερη επίσκεψη σας εκεί και τι πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν περισσότερο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο. Αυτή την ερώτηση έχουμε στην Ουγγαρία. Μάλιστα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και λιτά ευχαριστώ τον Επιτροπό για να μην αναλώσω άλλο χρόνο. Έκανε μια νομίζω εξαντλητική παρουσίαση, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσετε και να επιτηρήσετε την πλήρη υλοποίηση του ενεργειακού πακέτου μέτρων, γιατί είναι η βάση κίνησης για την δράση αυτή από σήμερα και όλα. Από την άλλη πλευρά απομένουν κάποια θέματα σημαντικά, πολλά από αυτά τα αναφέρατε. Αλλά ένα πρόβλημα που υπάρχει σε κάποιο βαθμό είναι ότι μπορεί να υπάρχει ο πειρασμός να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία θα γίνουν με με μονομένο τρόπο ξεχωριστά. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει να δω αν θα υποβάλει μια κοινή πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συνενώνει αυτές τις δράσεις όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα σε ένα ενιαίο πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε μια πλήρη επισκόπηση ας το πω έτσι αυτής της προσέγγισης για το ποια θα είναι αυτή η δράση, τα μέτρα αυτής της δράσης από τα θεσμικά όργανα και τελευταίο και πιο εξειδικευμένο ακόμα υπό τους όρους των επενδύσεων που θα χρειαστούν για την επένδυση στις επενδύσεις σε αυτά τα θέματα τα ενεργειακά. Πώς προβλέπετε ότι θα εγγυηθεί η πρόσθετη αναγκαία χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες αυτές χαμηλών εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα και χρήσης, ε, χρήση μειωμένης χρήσης του άνθρακα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φον Μπρέντ παρακαλώ. Ehm, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα είχα. Καταρχήν για το εγχείρημα αυτό της, στη Βόρεια ε, Θάλασσα υπάρχουν ε, μεγάλα προγράμματα offshore εγχειρήματα για την αιωλική ενέργεια. Είναι σημαντικό να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα προωθήσει. Θα ήθελα και θα ευχόμουν να γίνουν και περισσότερα πράγματα ακόμα. Πόσα κονδύλια μπορούν να διατεθούν ώστε να υπάρχει ένα ε, μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα σε τέτοια διαδικτύωση για αυτά τα δίκτυα offshore, παράκτια και ποια νομοθεσία χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά σε καλή νομοθετική βάση. Και δεύτερον, όσον αφορά την πυρηνική, τον ε, κύριο πυρήνα για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις που γίνονται θα πρέπει να μεριμνήσει η κοινότητά μας, η ευρωπαϊκή κοινότητα, να διασφαλίσουμε τα θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ραδιοπυρηνικά, τα πυρηνικά απόβλητα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ποια νέα στοιχεία υπάρχουν στη νέα πρόταση. Ο συνάδελφος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο κύριος Φλόρενς έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Επίτροπε, ακούω πάρα πολλά κατά καιρού για την ασφάλεια των ενεργειακών θεμάτων σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις, ε, την εκμετάλλευση του άνθρακα χαμηλών εκπομπών ρήπων. Και αν σκεφτεί κανείς ε, όλα αυτά, πώς μπορείτε να φανταστείτε ότι η ενεργειακή ασφάλεια με σταθερή και μεγάλη οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παλ Ρούιμπιχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά. Πρώτη ερώτηση. <clears throat> για μια ενιαία εσωτερική αγορά. Αν την θέλουμε, χρειαζόνται οι προϋποθέσεις για να την πετύχουμε. Κοινέ προκηρύξεις, δημόσιες προκηρύξεις ε, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες, παράδειγμα. Επόμενο βήμα πρέπει να είναι οι διαδικασίες αδειοδότησης, που και αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Ιδιαίτερα αδειοδοτήσεις <clears throat> που θα βρίσκονται υπό το πρίσμα του κοινού συμφέροντος, της κοινή ωφέλεια και τα ενεργειακά προγράμματα χαρακτηρίζονται από την κοινή ωφέλεια. Θα πρότεινα <clears throat> μια ομάδα εργασίας να δημιουργηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα ενέργειας αλλά και για τα θέματα περιβάλλοντος και με άλλους που θα εμπλέκονται και που με θετικό τρόπο θα αναπτύξει προϋποθέσεις για τις διατάξεις για την αδειοδότηση. Νομίζω θα ήταν πολύ επικοδομητικό για τα κράτη-μέλη να έχουν ένα τέτοιο πρότυπο. Πώς αποτελεσματικά και γοργά μπορούν να, να διευθετούνται, να ρυθμίζονται τα θέματα αδειοδοτήσεων, ώστε τα προγράμματα δράσης να μπορέσουν έγκαιρα να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με μια δεσμευτική πρόταση για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλας έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά τη δυνατότητα επίτευξης των δεσμευτικών εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περίοδους οικονομικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα φιλόδοξο δεσμευτικό στόχο για μερίδιο 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί εντατικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει το γενικό στόχο 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Οι στόχοι αυτοί υποτίθεται ότι πρέπει να επιτευχθούν παρά τις τεταμένες οικονομικές συνθήκες, διότι η πράσινη ανάπτυξη θεωρείται ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Πιστεύετε ότι αυτή η φιλόδοξη στόχη είναι πραγματικά εφικτή από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και ανέμε πιο κόστος για τη συνολική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Ζαντό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τον κύριο Αλμούνια, τον συνάδελφό σα, τον είχαμε ρωτήσει για τις κρατικέ επιδοτήσει προς τον άνθρακα. Και είχαμε πάρει μία απάντηση, ιδίω για την Ισπανία, που είχε δώσει μια, έναν ορίζοντα για το 2010 για να θεώρησε για αυτές τις κρατικές επιχορηγήσεις για τον άνθρακα. Εσείς πώς σκοπεύετε να τις χειριστείτε αυτές τις βοήθειες. Θα τις εγκαταλείψουμε λόγω των περιβαλλοντικών προκλήσεων που συνεπάγονται. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Συζητήσαμε με το Γενικό σας Διευθυντή για την ενεργειακή αποδοτικότητα ξαναείδε τους δεσμευτικούς στόχους στο επίπεδο των διάφορων ε, προϊόντων που έχουν σχέση με τον οικολογικό σχεδιασμό. Διότι είδαμε ότι το συνολικό ποσό όλων αυτών των ρυθμίσεων δεν επιτρέπει 20% εξοικονόμηση ενέργειας ως το 2020. Εσείς τι γνώμη έχετε βάσει των σημερινών αξιολογήσεων. Τι δεσμευτικό συνολικό στόχος μας χρειάζεται για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι, συνάδελφος παρακαλώ. Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στην ακρόαση συνέβη το εξή. Μία ερώτηση τίθετο, ακολουθούσε μία απάντηση. Τώρα είναι τόσες πολλές οι ερωτήσεις, τόσες ερωτήσεις, τώρα θα μπορέσουν να απαντηθούν. Δεν ξέρω. Τώρα, για την χρηματοδότηση, οδικοί χάρτες και τα λοιπά. Τι γίνεται, πώς μπορείτε για παράδειγμα, να τα χρηματοδοτήσετε όλα αυτά, ώστε να έχουμε αποκεντρωμένη, αποκεντρωμένο πλαίσιο διαμόρφωσης των ευθυνών και έτσι να λειτουργήσουμε. Να μπορεί και κεντρικά να δίνει εντολές και προς προσανατολισμούς η Ευρώπη, αλλά να έχουμε και το θέμα των εθνικών ευθυνών. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερο κάτι για τις απόψεις σας για τη χρηματοδότηση και τους οδικούς χάρτες και τα 500 εκατομμύρια για τους ε, ε, δήμαρχους και τους δήμους και τις κοινότητες σίγουρα θα χαίρονται οι δήμαρχοι γι' αυτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. κύριε Πίτροπε, κάποιες ερωτήσεις έχω για την Ουκρανία πρώτον. Ο πρόεδρος Πούτιν, λέει ο κύριος Μπιουτικόφερ, είπε ότι θα πρέπει να συγχωνευτούν οι μεγάλες επιχειρήσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Ε, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόταση κοινού κονσόρτσιου. Δεύτερον, είπατε, διμερείς πολιτικές ε, για τα ενεργειακά θέματα ας είναι παρελθόν. Η Αυστρία με το South Stream κάτι τέτοιο όμως συμφώνησε τώρα πρόσφατα. Μπορείτε να δώσετε μια υπόσχεση ότι δεν το βρίσκεται καλό αυτό και ότι κάτι θα κάνετε στο μέλλον να αποφευθεί αυτή, αυτή η πολιτική. Τρίτον, Ναμπούκο. Το, ο Ναμπούκο βρίσκεται επί ξηρού ακμής αυτή τη στιγμή και αν το Ναμπούκο δεν υλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους θα είναι παρελθόν, θα έχει πλέον ε, ιστορικό χαρακτήρα μόνο. Ποια είναι η, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά ε, των προθέσεων της Ιταλίας ή Γαλλίας να μπορέσει πραγματικά δεσμευτικά να προχωρήσει μέχρι τέλη του έτους ε, το Ναμπούκο. Είτε τώρα το κόστος εκρήγνεται. Γίνεται λόγος τώρα ότι πιθανώς ε, θα πρέπει να αναλάβουν πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αληθεύει αυτό. Πώς θα αποφύγετε περαιτέρω έκρηξη κόστους Υπάρχει ένας μηχανισμός ε, στον προϋπολογισμό για τη γεωργία που τον εφαρμόζουμε όταν υπάρχει έκρηξη κόστους. Θα χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο μηχανισμό και για το ΙΤΕΡ. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση ο κύριος Μέτεχάους παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε ο κύριος Μέζαρος. Χαίρομαι για το ότι αρκετοί έθεσαν το ε, θέμα αυτό. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει και εμείς να το αναφέρουμε. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τελική ρύθμιση αυτού του θέματος διότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα της αλλαγής ε, της των κλιματικών αλλαγών Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μια συμφωνία. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες ε, δεν μπορούν να διασφαλιστούν ε, χωρίς ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας. Με το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων και χωρίς συγκεκριμένες προοπτικές δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι 40% των εκπομπών ρήπων ε, προκαλείται από τις οικοδομικές αυτές δραστηριότητες. Ποια είναι η άποψή σας για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Έχετε κάποια άποψη. Ντί παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για το ότι ήρθατε εδώ πέρα, γιατί δείχνετε ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις υποσχέσεις σας. Παγκόσμιο ζήτημα η ενέργεια και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις. Ποια είναι η άποψή σα για την πορεία της ενέργειας παγκοσμίω και τα όσα έγιναν στην Κοπενχάγη που έχουν να κάνουν με την ενέργεια της κλιματικές αλλαγές μπορούν να αλλάξουν την άποψή σα. Αύριο θα έχουμε, μεθαύριο μάλλον, τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς εξελίσσεται ο διατλαντικός διάλογος για τα ζητήματα αυτά και πιο συγκεκριμένα για την πυρηνική ενέργεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να αποθηκεύονται με συγκεκριμένο τρόπο τα πυρηνικά απόβλητα, ενώ άλλα κράτη-μέλη όπως η Γαλλία προτιμούν την ανακύκλωσή τους και όχι την αποθήκευση. Και επίσης, ποια είναι η θέση όσον αφορά το ίτερ πέρα από τα χρηματοδοτικά ζητήματα. Υποστηρίζετε εσείς το πρόγραμμα ίτερ και θα μπορούσατε επίσης ε, να μας πείτε πώς προγορά το TESERTEC, δηλαδή η ε, ενέργεια μέσω των ηλιακών πάνελ ε, στην έρημο στο Μαγκρέμπ. Κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Υπακούντα τον Επίτροπο, δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη. Εσείς αναφέρατε <clears throat> το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης και πόσο σημαντική είναι. Ερώτησή μου. Έλαβε απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> για το πώς θα υπάρξει διευκόλυνση πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και τι θα γίνει με αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Εν ώψη της εκκίνησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας πρότασης για ένα νέο πακέτο για ενεργειακές υποδομές, ποια μέτρα σκέπτεστε να προτείνετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βέμπερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε, κύριε Επίτροπε, ότι θα προβλέψετε δρακόντια μέτρα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Την υπερθέρμανση δηλαδή του πλανήτη. Ε, μιλήσατε εδώ για την ε, οικοδόμηση εκτηρίων, την κατασκευαστική δραστηριότητα που δεν σέβεται αυτού του κανόνε πλήρω. Το θέμα είναι λοιπόν πώ θα ισχύουν, ποια θα είναι τα κριτήρια και ποιο ο τρόπο ελέγχου υλοποίηση των κανόνων. Τι διαθέτετε και τι σκοπεύετε να προβλέψετε. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωση υπάρχουν ρυθμίσει και κανόνε σωρό, αλλά πολλές φορές η έλεγχη στην πράξη είναι πολύ λίγο αποτελεσματική, για να μην πω καθόλου. Έτσι λοιπόν, κανόνε χωρί ε, περαιτέρω ελέγχου για να δούμε τι γίνεται στην πράξη, συχνά είναι μόνο λόγια στο χαρτί. Ποια θα είναι τα μέσα ελέγχου που ήδη διαθέτεται και θα προβλέψετε, για να είσαστε βέβαιοι ότι θα τηρηθούν οι κανόνε που εμεί υπαγορεύουμε. Η συνάδελφος Μέρκης η επόμενη, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μία ερώτηση έχω. Ουσιαστικά δύο. Κάνατε λόγο για μεγάλα προγράμματα, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είπατε. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Τα άλλα 20% όσον αφορά τη μείωση των, ε, ε, της πατάλης ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τι εννοείται ακριβώς, ποια συγκεκριμένα μέτρα έχετε υπόψη σας να λάβετε. Και έχω και μία ακόμα ερώτηση. Βρίσκω τα μεγάλα προγράμματα, όπως όλοι, πολύ ωραία. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα να υιοθετούμε μικρά προγράμματα και να τα προχωράμε. Και έτσι μπορεί κάτι να γίνει για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και της ενεργειακής αποδοτικότητας και της στρατηγικής για το 2020 2020 στους στόχους μας. Και εδώ η ερώτηση, πώς βλέπετε εσείς υπάρχει μια δυνατότητα με μικρά προγράμματα και εγχειρήματα να ξεκινήσουμε για πολίτες για παράδειγμα να κινητοποιηθούν να υπάρχει ενεργειακή αποδοτικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρο, για παράδειγμα ε, γεννήτρες, μικρογενεά προγραμμάτων. Η κυρία Φιγερέδο παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Απλά και μόνο μία ερώτηση κύριε Επίτροπε. Είμαστε στο ευρωπαϊκό έτος της καταπολέμησης της φτώχειας και όταν δούμε μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση των ατόμων, των ανθρώπων σε είδη πρώτης ανάγκης και βλέπουμε το βαθμό στέρησης, για παράδειγμα, των πολιτών όσον αφορά αυτά, όσον αφορά τη θέρμανση των σπιτιών τους, για παράδειγμα. Τι βλέπουμε. Διαπιστώνουμε ότι σε διάφορες χώρες το ποσοστό της στέρησης ε, θέρμανσης των ε, κτηρίων, των σπιτιών είναι ανώτερο ποσοστό από 30%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια φτώχεια ενεργειακή σήμερα. Ενεργειακή όσον αφορά την πρόσβαση σε ε, ε, τέτοιες πηγές ενέργειας για τη θέρμανση για τους πολίτες μας. Σας ερωτώ για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακολουθείτε. Έχετε κάποια πρόταση για να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ως ένα ορόσημο κιόλα, ω ένα σημείο τη καταπολέμησης τη φτώχεια στο, ενεργεια, στο ευρωπαϊκό αυτό έτος. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Όλες οι ερωτήσει καλύφθηκαν. Τώρα έχει ο Επίτροπος την ευκαιρία αυτές τι πολλές ερωτήσεις να τις απαντήσει σε λεπτομέρειε. κατά λεπτό. Έχετε τον λόγο, Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, το Nord Stream ήταν η πρώτη ερώτηση που μου θέσατε. Πιστεύω ότι στην ιστορία γενέσεως το Nord Stream δεν ήταν ένα ευρωπαϊκό καθαρά πρόγραμμα. Έγινε ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποδομών με ιδιωτικές συμβάσεις. Τα όμορα κράτη, τα γειτονικά κράτη έδωσαν άδειε σε σχέση με τις ε, ε, δεσμεύσεις τους ε, για την προστασία του περιβάλλοντο και σε σχέση με την ε, ε, εκτέλεση του προγράμματος αυτού. Βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτό. Και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δεν είναι μειονέκτημα, αλλά πλέονέκτημα. Τεχνικά, τεχνολογικά, ακόμα και αν όσον αφορά τη χώρα προέλευσης ε, για το φυσικό αέριο δεν θα είναι ασφάλεια. Όμως το Ναμπούκο θα ήταν διπλά αξιόλογο. Πρώτον τεχνικά, τεχνολογικά και δεύτερον όσον αφορά την προέλευση του φυσικού αερίου που θα μας έδινε ασφάλεια. Και πρέπει να δούμε την ε, ε, εφέτος και το βλέπουμε αυτό ανάγλυφα. Σύντομα θα σας το αναφέρω. Είχα πάει στο Ασχαμπάντ και είναι πρόθυμοι εκεί να δώσουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια συμβάσεις για παροχή φυσικού αερίου. 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τους ε, κύκλους της κυβέρνησης που λένε μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο, μία υπογραφή, μία εγγύηση. Το καλύτερο θα ήταν ο Μπαρόζο να υπέγραφε. Δεν είναι πολύ απλό στους τουρκμένους εταίρους μας να εξηγήσουμε ότι ένα κονσόρσιο φυσικού αερίου από την ΕΡΒΕ και άλλες εταιρείες αποτελείται. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπογράφει εκείνη, δεν είναι κεντρικό κράτος όπου υπάρχει αυτή η υποχρέωση δέσμευσής του. Δηλαδή η, υποχρέ... η εγγύηση της αγοράς φυσικού αερίου σε προσιτές τιμές είναι σημαντικό θέμα. Σε σχέση τώρα με το ίδιο το πεδίο ε, κοιτασμάτων φυσικού αερίου φαίνεται ότι μπορεί να είναι εφικτό αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει εδώ και η BP και η Total που είναι πρόθυμοι για την ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κασπία θάλασσα 20 δις ευρώ να διαθέσουν, 20 δις ευρώ ώστε αυτό το αέριο να αντληθεί. <clears throat> Τρίτον, ένα ανοιχτό θέμα είναι η μεταφορά φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν ως τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. <clears throat> Μια, η τουρκμενική κυβέρνηση θα προτιμούσε με πλοία να μεταφέρεται. Μειονέκτημα, πανάκριβη αυτή η μεταφορά. Και δεν είναι ακόμα απόλυτα αποδεδειγμένη η, η βιωσιμότητα αυτού. Έχουμε και το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου. Έχουμε θέματα διεθνούς δικαίου. Είναι λίμνη ή Κασπία θάλασσα ή θάλασσα. Και έχουμε εδώ και θέματα που ε, εμπλέκουν και αφορούν ίσως και τη Ρωσία σχετικά. Τον Μπακού πιέζει να ληφθεί απόφαση εφέτος και για την παροχή σταθερά 17 ε, ε, δισεκατομμυρίων κυβικών ε, μέτρων φυσικού αερίου ετήσια. Παρόλα αυτά, οι, οι Ρώσοι πιέζουν να μην γίνει αυτό. Οι Ρώσοι λένε ότι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται από την Κασπία στη Ρωσία. Η δική μου προσέγγιση είναι διαφορετική. Οι Ευρωπαίοι τώρα θα πρέπει να δουν και την δυνατότητα εμπλοκής και των Κινέζων και μεταφορά προς την Κίνα. Έχουμε εδώ ένα, ας το πω, μια πλατφόρμα και παίζει το Αζερμπαϊτζάν στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη, ας το πω έτσι. Θα φτάσει αυτό το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Από αυτές τις αποφάσεις εξαρτάται. Οι Κινέζοι όμως είναι ταχύτεροι από ό,τι μπορεί κανείς να υποθέσει. Και το θέμα της διάβασης μέσω από τη Γεωργία είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής που εμπλέκονται. Η συμφωνία Αζερβαϊζάν-Τουρκίας είναι σημαντική. Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε καλή πορεία. Έχω υπόψη να πάω ε, και στην Άγκυρα και τα κράτη-μέλη πρέπει όλα, όλα να δώσουν την αναγκαία αυτή δέσμευση την οποία έδωσαν να την τηρήσουν, με συγχωρείτε, να τηρήσουν αυτή τη δέσμευση. Όλα και η Αυστρία. Αν παράλληλα τώρα με το South Stream θα προχωρήσουν τα έργα, ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε. Παρόλα αυτά όμως η δέσμευση ότι η ευρωπαϊκή υποδομή θα μπορέσει να καταστήσει εφικτό τον Αμπούκο είναι σημαντικό και θα πρέπει να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε Σωστά είπατε, τα 30% ίδια κεφάλαια, να διασφαλιστεί το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων. Και για το 70% με συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δούμε πώς μπορούν οι πιστώσεις να διατεθούν. Τελευταίο σημείο. Απομένει αυτή τη στιγμή στην αγορά φυσικού αερίου ε, απομένουν δύο παράγοντες ανασφάλειας, αβεβαιότητας. Είναι μικρότερη η ανάγκη σήμερα από ότι αυτή που είχε προβλεφθεί πριν από τρία χρόνια. Και τα νέα κοιτάσματα και η εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων δημιουργούν ξαφνικά, ας το πω έτσι, μια αβεβαιότητα για την σημασία των αγωγών φυσικού αερίου και των, της κεντρικής παροχής ε, φυσικού αερίου που μέχρι στιγμής ε, δεν είχε ε, διασφαλιστεί. Και <clears throat> το liquid gas, το ρευστοποιημένο φυσικό αέριο, είναι και αυτό σημαντική υπόθεση. Τώρα, για το το θέμα του άνθρακα και το πώς θα αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω ότι μακροπρόθεσμα παγκόσμια ο άνθρακας θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο στην Κίνα, στη Ρωσία, στη ΣΥΠΑ. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί σημαντικό ρόλο έχει ο άνθρακας. Στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες ε, πάλι υπάρχει και το θέμα του άνθρακα. Γι' αυτό λέμε ότι σε μείγμα ενεργειακό <clears throat> οι αντιδραστήρες, οι μονάδες που καίνε άνθρακα θα διαδραματίσουν ένα ρόλο και θα πρέπει εδώ να δούμε τι θα γίνει με τη σύλληψη και την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι βέβαιο και δεν έχω σαφή απάντηση ποιες τεχνολογικές δυνατότητες θα είναι εφικτές στο μέλλον. Όσον αφορά την καινοτομία για παράδειγμα, η δική μου τοποθέτηση αφορούσε ένα και μόνο πρόβλημα. Όχι σε σχέση με το ε, Βραδεμβούργο και την ε, εκμετάλλευση του, την χρήση του ε, άνθρακα, παράλληλα με άλλες, άλλα τέτοια εγχειρήματα. Και για το ότι θεωρώ δύσκολο να υλοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Αν δούμε τώρα τις δημόσιες τοποθετήσεις και σε σχέση με τη Βουλή μας, παραγωγή για παράδειγμα στην περιοχή του Ρούρ και όλα αυτά θέτουν δυσχέρειες. Η δική μου τοποθέτηση αφορούσε το ποιος θα αναλάμβανε αυτή την επιβάρηση και ότι θα έπρεπε να υπάρχει αντιστάθμιση οικονομική. Και αυτό είναι κάτι το πρωτοπόρο, διότι και η επιβάρηση στις υποδομές, ακόμα για παράδειγμα και για τη χρήση ε, αντισταθμιστικά κάποιων δικτύων, θα πρέπει να δούμε και τις ε, κοινωνικές ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνονται και την αλληλεγγύη που πρέπει να εκφράζουμε. Γι' αυτό, σε αυτό αναφερόταν η τοποθέτησή μου για το πρόγραμμα αυτό, για την έρευνα σε ανταγωνισμό και με άλλες χώρες παγκόσμια, που θεωρώ ότι παραμένει αναλύωτο και έχει μεγάλη προτεραιότητα. Εσείς, ε, κύριε Ευρωβουλευτά, θέσατε το ερώτημα <clears throat> τι θα γίνει με την απελευθέρωση κονδυλίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε η προηγούμενη Επιτροπή στην κρίση, ένα δις για να δοθεί ανακούφιση στα, στις περιοχές που πλήττονται από την κρίση. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο 100% μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τα περισσότερα κονδύλια αντλήθηκαν, αλλά δεν έχουμε όλα τα προγράμματα τα οποία να έχουν υλοποιηθεί. Απομένουν κάποια ποσά και θα δούμε ότι σε 8 εβδομάδες θα γνωρίζουμε περισσότερα για το ποια κονδύλια δεν θα έχουν ε, καταβληθεί. Και τότε θα έχουμε περίπου 115 εκατομμύρια. Αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς ε, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Φανίστερ Ρόι, μπορούν ίσως να υπάρξουν τα 500 αυτά, αλλά τουλάχιστον 115 αυτή τη στιγμή. Τώρα, ποιο θα είναι το τελικό ποσό θα το ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες. Και αυτό είναι σημαντικό αν θα ξέραμε ε, μετά από ένα εξάμεινο θα ήταν πολύ καθυστερημένη η χρονική στιγμή για να δράσουμε. Πρέπει να βρούμε ένα χρονικό σημείο Ιούνιο-Ιούλιο για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε περίπου ποια θα είναι τα απελευθερωμένα αυτά κονδύλια που θα διατεθούν ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ώστε οι στόχοι που επιθυμείτε εσείς, αποδοτικότητα στην ενέργεια, να μπορέσουν να ε, καλυφθούν, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν έτσι και εργαζόμαστε ώστε πριν από τις θερινές διακοπές να καταφέρουμε σε ένα παράθυρο ευκαιρίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πούμε και να κρίνουμε τόσα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Tech είναι ένα πρόγραμμα για την ε, ηλιακή ενέργεια και την ε, αιωλική ενέργεια και όχι για φυσικό αέριο ή άλλες ε, πηγές ενέργειας. Και γι' αυτό για μας ε, η υποστήριξη του ΝΤΕΖΕΤΕΚ έχει αποφασιστική σημασία και θα εξαρτάται όπως και σε σχέση με τα ε, θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποθέτω ότι παρόλα αυτά για τις υποδομές, τη χρηματοδότηση δηλαδή των γραμμών και των δικτύων, θα πρέπει να υπάρξουν ενισχύσεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μία θα μπορούσα να φανταστώ, δηλαδή την ε, διασφάλιση ενεργειακών πόρων ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαχάρα, ώστε μακροπρόθεσμα να υπάρχει εγγύηση διασφάλισης ενός συγκεκριμένου ποσού μιας για την τιμή αυτού του ε, προϊόντος της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κάτι που στην ε, Γερμανία με αυτόν τον τρόπο θα ήταν βιώσιμο. Αξίζει να το συζητήσουμε υπό την πτυχή της ενεργειακής ασφάλειας. Για τους ε, οδικούς χάρτες 2050 δεν είμαστε εμείς ε, δούλοι κάποιων καθηγητών και υπήκοοι τους, δεν ξέρω καν αυτόν τον κύριο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, μελέτες που μπορεί κανείς να ε, λάβει υπόψη του. Έχουμε και ότι από μια μελέτη ότι 80% και παραπάνω είναι εφικτό. Και όλα αυτά γίνονται υπό συγκεκριμένε προοπτικέ. Θα λάβουμε υπόψη και θα προσπαθήσουμε να δούμε με τη μέγιστη αντικειμενικότητα τι μπορεί να γίνει. Και μάλιστα είναι ένα πρόγραμμα, θα έλεγε κανεί ε, ολόκληρου αιώνα δράσεων. Μιας ολόκληρης πεντηκονταετία τουλάχιστον. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν έχω δεσμευτεί ακόμα, δεν έχω καθορίσει και δεν έχω δεσμευτεί συγγνώμη, πρέπει να σέβομαι αυτά που κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό που κάνει ο Γιούνκερ, αυτά που κάνουν οι αρχηγοί κρατών, ναι, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τεχνικά, οικονομικά για μια χώρα είναι κάτι εφικτό ή όχι και να αποφασίσουμε από κοινού πώς μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέχρι το 2050 θα πορευτούμε. Μετά είχαμε το θέμα της ε, ε, εκμετάλλευσης ε, της ε, υδάτινης ενέργειας. Ε, έχουμε το θέμα που πρέπει εδώ να δούμε από κοινού, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τότε βιώσιμη όταν από πλευράς δυναμικού και αποθήκευσης προϊόντος μπορεί να προχωρήσουμε. Η υδροηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει ρόλο εδώ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επίσης. Οι συσσωρευτές, οι μπαταρίες, είναι σαφές όμως ότι σήμερα σε σχέση με την αποθήκευση δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Πολύ απέχουμε μεγαλύτερη αποθήκευση ε, υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί και εύκολα κιόλας ε, στην Ευρώπη. Διότι στο τέλος τέλος η αποδοχή επιτόπου από τους πολίτες, τουλάχιστον σε περιοχές όπου βρίσκονται πυκνοκατοικημένες πόλεις ε, ή στις Άλπεις για παράδειγμα όπου έχουμε το θέμα της προστασίας της φύσης θα υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις. Το 8ο πρόγραμμα έρευνας τώρα για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Έχω λιγότερη πείρα σχετικά με σας. Πρόκειται για το θέμα ποια είναι η σημασία της έρευνας τα επόμενα χρόνια, τα οικονομικά αυτά χρόνια. Στο Κοινοβούλιο σε εσά, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε την ε, θεματοποίηση αυτών. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό για την γεωργία, για τα περιφερειακά προγράμματα, για την έρευνα επίσης. Προετοιμασία προϋπολογισμού. Μετά έχουμε το θέμα τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη και τι θα δώσουν. Θα παραμείνουμε στο 1, τόσο του ΑΕΠ ως μέρος ενός ΑΕΠ που έχει ήδη μειωθεί κατά 4% σε πολλές χώρες. Το 2030 θα έχουμε μικρότερο ποσό ίσως από ε, κάποιο οικονομικό έτος λόγω της ε, μείωσης ε, του ε, ΑΕΠ. Θα δεχθούμε την οροφή ή θα, θα ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια για περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει κάθε ένας από εμά με την κυβέρνησή του και το κόμμα του στη χώρα του να τα συζητήσει στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών εξίσου. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε εσείς στις χώρες σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η κοινή επιτυχία μας. Αυτή είναι η ανάγκη έτσι να προχωρήσουμε. Και όταν θα ξέρουμε τι θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρώπης συνολικά, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι θα διατεθεί στην έρευνα. Έχουμε συζητήσει σε σχέση με την Επίτροπο για την έρευνα και τους αρμόδιους συναρμόδιους για τα θέματα αυτά θα προσπαθήσω να δώσω μάχη για να δοθούν το δυνατόν περισσότερα κονδύλια στην έρευνα. Και μετά θα συζητήσουμε τι θα γίνει με τα τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή οικονομία, ώστε να πετύχουμε με το ένα ευρώ που διαθέτουμε περισσότερο από ένα κανονικό άλλο εγχείρημα με ένα ευρώ που για κάθε ευρώ να υπάρχει υπεραξία. Και θα έχουμε και ε, σε σχέση με τις ε, αποφάσεις στη Λιουμπιάνα για παράδειγμα να υπάρξει η, δυνατότητα να είμαστε παρόντες ώστε αυτή η ρυθμιστική αρχή, αυτή η υπηρεσία να είναι έτοιμη να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να μπορέσει η ολοκλήρωση, ο εναρμονισμός των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να επιτευχθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο καλύτερα. Και μετά είχαμε και το θέμα του ΙΤΕΡ. Το ΙΤΕΡ τι είναι είναι ένα παιδί το οποίο υιοθέτησα εγώ, το παρέλαβα από άλλον. Είναι, είχαμε και κάποιες αρνητικές εξελίξεις. Η πρώτη αρνητική εξέλιξη, όπως πολλά δημόσια προγράμματα, <clears throat> έχουμε εδώ το κόστος που είχε υποβαθμιστεί, είχε υποτιμηθεί. Το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε προϋπολογιστεί. Δεύτερον, οι ο, κατευθύνσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτω από το ευκταίο τα, οι επιδόσεις. Τρίτον, οι οικονομικοί κύκλοι δεν συμμετείχαν επαρκώς όπως θα έπρεπε. Τέταρτον, οι εταίροι, ιδίω η ΕΠΑ, την δική μας αυτή συνεμπλοκή, την ε, ε, αναμένουν. Όμως ε, αναμένουν οι εταίροι να κάνουμε περαιτέρω λάθη εμείς ή να μην τα πάμε όπως θα έπρεπε καλά. Και τότε η ευρωπαϊκή ή η γαλλική ηγεσία σε αυτά τα θέματα όπου συμμετείχαν για παράδειγμα οι άλλοι θα συρρυκνωθεί. Και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό ε, το ε, εγχείρημα. Θα παρουσιαστεί έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε καλύτερες επιδόσεις. Πρόκειται ε, για ε, δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Σας λέω ειλικρινά, θα βάλω τα χαρτιά στο τραπέζι, διότι η σαλαμοποίηση, η, η κατατμημένη πολιτική δεν οδηγεί πουθενά και είναι η λάθος πολιτική παγκοσμιοποιημένα. Πρέπει να είναι σαφές όμως, αν το ίτερ από τους ίδιους τους Ευρωπαίους στριμωχθεί και κολλήσει στον τοίχο, τότε η ΙΠΑ, οι Ινδίες, η Ινδία και η Κίνα με κανένα πρόγραμμα, σε κανένα τομέα δεν θα θέλουν να είναι οι Ευρωπαίοι οι πρωτοπόροι και οι επικεφαλείς. Πρόκειται για το ίτερ και για παραπάνω θέματα, για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μεγάλα κράτη-μέλη στην παγκόσμια έρευνα να είναι πιστικά και να μπορούν να αναλάβουν ένα ηγετικό ρόλο. Αυτή είναι η λιδία λίθος η δοκιμασία εδώ. Μετά είχαμε και το ερώτημα πώς τα αιωλικά ε, παράκτια κέντρα θα τα προωθήσουμε στη Βόρεια Θάλασσα. Στο πρόγραμμα των υποδομών έχουμε προβλέψει τέτοιες δράσεις. Παρακολουθούμε αυτό το εγχείρημα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως εγώ είμαι πεισμένος ότι πρωτογενώς πρέπει να είναι αυτά αποδοτικά. Για παράδειγμα, θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σημαντικό κονδύλιο για τις αναγκαίες δράσεις. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί, για παράδειγμα, δύο-τρία 4% συμπληρωματικά να διαθέτει. Όμως το κύριο έργο θα παραμένει έργο των οικονομικών κύκλων, των εταιριών, των εταιριών ενεργειακών προϊόντων, ώστε εκείνοι να μπορούν να συμμετέχουν. Το σημαντικότερο έργο της αρχής των, ε, των ρυθμιστικών αρχών είναι να υλοποιηθεί αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μια συμπληρωματική διάσταση από πλευράς χρηματοδότησης της Ευρώπης, ναι, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε την κύρια ευθύνη για αυτές τις τεράστιες επενδύσεις ο κύριος Ρούμπιχ ρώτησε αν για αδειοδοτικά θέματα, για υποδομές, για θέματα υποδομών, για τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις ε, κάτι μπορεί να γίνει ευρωπαϊκά. Ο κώδικας βέλτιστων πρακτικών θα έλεγα εδώ πρέπει να ακολουθηθεί γιατί κατά τα άλλα είναι σαφές όσον αφορά το πρόγραμμα και την έγκριση των αδειών και την αδειοδότηση ακόμα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα εξακολουθήσει να, παραμένει, εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πώς θα πετύχουμε τον στόχο 20-20-20, πολύ θεμητή και δικαιολογημένη ερώτηση. Δεν θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας ε, και να περιμένουμε μέχρι το 2015 και τότε να πούμε κάτι χάσαμε την ευκαιρία τη χρονική να δράσουμε. Διαπιστώνω αναλύωτα και μέσα σε συγκυρία κρίσης ότι η μεγάλη αποδοχή υπάρχει από τους πολίτες για το 2020-2020 στην οικονομία, στην πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης, στην επιστήμη, από τους επιστημονικούς κύκλους. Δεν διαμφισβητούνται αυτά. Δεν ξέρω πολλά τέτοια στοιχεία που να είναι τόσο αποδεκτά από τους πολίτες και να έχουν τέτοια αποδεκτικότητα όπως αυτή η στοχη 2020 20-20-20. χωρις μικρόφωνο η παρέμβαση, δεν ακούγεται. Δεν το, δεν το πιστεύω θα λέγα αυτό. Μην ανησυχείτε. Θα έχω, θα έχω επαφή κατηδίαν μαζί του. Υπάρχει πολύ μεγάλη αποδεκτικότητα λοιπόν, αποδοχή όλων αυτών. Και αν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να κάνουμε τον εξή, να ακολουθήσουμε τον, κανένα, τον κανόνα όσο το δυνατόν λιγότερες περιοριστικές αριθμιστικές διατάξεις και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές διατάξεις. Και να μην χάσουμε το ε, χρονοδιάγραμμα, την ευκαιρία αυτή που θα μας δοθεί. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εθελοντική συμμετοχή από τους οικονομικούς κύκλους όσον αφορά τη συμμετοχή τους. Η Ουκρανία, κύριε Πιούτι Κόφερ, και εγώ το διάβασα αυτό που είπατε, αυτή την προσφορά μιας συμφωνίας Gazprom δηλαδή και της Ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου. Ο Ουκρανός Υπουργός είναι αυτή τη βδομάδα στις Βρυξέλλες, θα τον συναντήσω ε, δεν πρόκειται τώρα να υπάρξει κάποια δημόσια τέτοια δέσμευση, όμως είναι σαφές ότι η εταιρική σχέση με την Ουκρανία είναι τώρα κάτι που έχει οριμάσει για να συζητηθεί. Η νέα κυβέρνηση έχει την ε, δική μας εμπιστοσύνη, μια και δημοκρατικά εξελέγει και εκφράζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε κάποιες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή μια οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα επεβάρυνε αυτές τις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και δεν θα τις διευκόλυνε. Το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των κτηρίων μου φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ φλέγον θέμα. Και θα έλεγα ότι εμείς με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα το πεδίο των κτηρίων που ήδη υφίστανται έχουμε τεράστια δυνατότητα, μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ε, ενεργειακών πόρων. Πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε η εθνική εξυγίανση και τα προγράμματα ε, ε, εξυγχρονισμού και ανανέωσης ε, των κτηρίων επαρκούν ή πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να, είμαστε, έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα συζητήσω με τους αρμόδιους υπουργούς στα κράτη-μέλη και θα εξετάσω και θα δω ποια είναι η αποδεκτικότητα, η αποδοχή από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, αν ήταν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για τον Αντιπρόεδρο Biden, Biden τον είπα που θα έρθει ε, στις Βρυξέλλες και το θέμα της Κοπεχάγης θα πρέπει αντίστοιχα να συζητηθεί. Είναι η κυρία Χίλεγκαντ στην Βόνη και θα έχουμε και τη στρατηγική μας που θα καθορίσουμε για το Κανκούν. Διότι ήταν σαφές ότι η, Κοπενχάγη, η σύνοδος της Κοπενχάγης δεν ήταν επιτυχία για την Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρέθηκε σε εκείνα στο σημείο στο οποίο θα έπρεπε να έχει βρεθεί, δεν άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να μπορέσει να τεθεί στους Αμερικανούς το ερώτημα με το πετρέλαιο τι γίνεται. Η καταστροφή ε, στον κόλπο του Μεξικού δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι με επικίνδυνες τεχνολογίες να έχουμε το πετρέλαιο στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Και όχι μόνο το κλίμα, οι κλιματικές αλλαγές, η ίδια η φύση δεν μπορεί να υποτιμηθεί και έχουμε ε, βλάβες που είναι τεράστιες. Έχουμε εδώ Και το άλλο θέμα, το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Μια Ευρωβουλευτήνα ανέφερε αυτό το θέμα. Εγώ λέω ότι η Βελγική Προεδρία <clears throat> θα θέσει αυτό το κέντρο βάρους στις ε, ε, προτεραιότητές της. Παρότι οι εκλογές στο Βέλγιο δυσχεραίνουν και περιπλέκουν αυτό το θέμα, οι εκλογές στο Βέλγιο, το θέμα της Βελγικής Προεδρίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός ε, των ε, κυβερνήσεων που είναι ευάλωτες στα κράτη-μέλη είναι ένα πρόβλημα. ας αναμείνουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση των εκλογών στο Βέλγιο. Και για το θέμα της ενεργειακής φτώχεια θα το δούμε. Αναφέρεται από τη βελγική κυβέρνηση και εμεί θα ανταποκριθούμε σε αυτή την προτεραιότητα. Γι' αυτό το έργο θα πρέπει να δούμε να υπάρχουν προσιτές τιμές ενεργειακών προϊόντων, η εσωτερική αγορά, ο ανταγωνισμός, η ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Διότι κατά τα άλλα η ενεργειακή φτώχεια είναι μέρος, τμήμα της φτώχειας συνολικά και έτσι τμήμα, μέρος των εθνικών πολιτικών αναλύωτο παραμένει ότι πρώτα οι εθνικές πολιτικές ε, έναντι όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τίνει προς την διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρικοδοτώντας τις πολιτικές με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι με τα κοινωνικά μέτρα στο εθνικό επίπεδο να έχουν τα αναγκαία ενεργειακά προϊόντα σε προσιτές τιμές ώστε να μπορούν να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή με θερμενόμενη το χειμώνα πρέπει κατεπηγόντως ε, να αποχωρήσω. Έκανα ό,τι μπόρεσα να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Πρέπει να αποχωρήσω, να προσφωνήσω τους δημάρχους. Εκείνες ερωτήσει ερωτήσεις ε, που δεν έγινε δυνατό να τις καλύψουμε, να μου τις ξαναθέσετε και στο μέλλον ε, είμαι πρόθυμος να έχω και κατηδίαν επαφές μαζί σας. Σας ευχαριστώ όλους σας θερμά. Ευχαριστούμε Κύριε Επιτροπέ, νομίζω ότι ήσασταν διεξοδικό. Ε, καλύψατε σχεδόν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Όπω το είπατε και ο ίδιο, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε. Πρέπει όμω να φύγετε. Κανένα πρόβλημα. Σα ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό σημείο. Γι' αυτό θα ήμουν ευγνώμων. Αν όλοι οι φιλοξενούμενοι που εγκαταλείπουν την αίθουσα να την εγκαταλείψουν γοργά, σύντομα. Έχουμε ένα σημαντικό σημείο στην ημερησία διάταξη ακόμα. Είναι δυνατόν να φύγετε ήσυχα παρακαλώ και γρήγορα. Ήσυχα, χωρίς να κάνετε φασαρία και γρήγορα. Σημαντικό, έχουμε ακόμα ενδιαφέροντα σημεία που πρέπει να συζητήσουμε στην ημερησία διατάξη. Τώρα θα συζητήσουμε το θέμα της εντολής για την τριμερή, τον τριμερή διάλογο <clears throat> για το σχέδιο προϋπολογισμού 2011. Η συνάδελφος κυρία Edith Herzog είναι η συγγήτρια, έχει κάνει πολλή δουλειά για το θέμα. Είχαμε και μια εξαιρετική προσυζήτηση με τους ενδιαφερόμενους σκιώδεις εισηγητές και αυτό θα είναι επικοδομητικό τώρα για μας. Όμως πιέζει ο χρόνος τώρα στενά χρονικά όρια έχουμε και γι' αυτό θα πρέπει νυφάλια και ήρεμα να το ξανασυζητήσουμε. Η κυρία Χέρτσοκ θα έχει τον λόγο πρώτη όταν εγκαταλείψουν οι άλλοι την αίθουσα. Και με ησυχία παρακαλώ να φύγετε. Κυρία Χέρτσοκ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που παραμένουν στην αίθουσα γιατί βρίσκουν ενδιαφέρον το θέμα του προπολογισμού του 2011. Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Ήτρε το αργότερο στις 11 Μαΐου. Γι' αυτό και είχαμε έκτακτη συνεδρίαση της Ήτρε σε σχέση με τις τροποποιήσεις. Με τις τροπολογίες, συγγνώμη. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε να προλάβουμε και τις τροπολογίες ως τις 11 Μαΐου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, λοιπόν, για την Επιτροπή Ήτρε για το σχέδιο προπολογισμού 2011 είναι η 7η Μαΐου, η μαιου 7 Μαΐου το μεσημέρι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που είχα να αναγγείλω. Να πω όμως και λίγα λόγια για το λόγο που μας οδηγεί να εξετάσουμε με πολύ προσοχή και με ιδιαίτερη σοβαρότητα τον προπολογισμό του 2011. Δύο είναι βασικοί παράγοντες. Τον ένα τον ανέφερε ήδη και ο Επίτροπος, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο προπολογισμός του 2011 θα είναι κάπως πιο σφιχτός για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η διαδικασία προπολογισμού του 2011 είναι η πρώτη, η οποία βάσει τις συνθήκες της Λισαβόνας απαιτεί τη συμμετοχή μας. Είναι ευκαιρία να αναλάβουμε πλήρως τα καθήκοντά μας. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ήτρε, διότι μεταξύ των προεδρετήτων της Ήτρε, όπως οι ενεργειακές επενδύσεις, η χρηματοδότηση του νέου διαστημικού χώρου, των πολιτικών καινοτομιών και των ε, ερευνητικών πολιτικών είναι όλα αυτά νέα στοιχεία σε σχέση με τον προπολογισμό του 2010. Οι αρμοδιότητέ μα λοιπόν ε, εμπλουτίζονται. Ενώ ο προπολογισμό όμω τη Ευρωπαϊκή Ένωση συρρυκνώνεται. Πρέπει λοιπόν ω το δυνατόν περισσότερο να είμαστε ενωμένοι αν θέλουμε να έχουμε περισσότερα επιτεύγματα. Τώρα από την δημοσιονομική την άποψη. Πώ έχει ο προπολογισμό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι λόγω τη οικονομική κρίση και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και των οικονομικών του πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική από την προηγουμένως, αλλά μας περιορίζει και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο ήδη έχει δείξει ότι ε, παρουσιάζει ελλείψεις για την ε, χρηματοδότηση βασικών προγραμμάτων όπως τον Καλλιλέο, το GMS, ε, το πρόγραμμα της κοινωνικής ένταξης, του επισητισμού για τις φτωχότερες χώρες ή του προγράμματος ανάκαψης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να καλύψουμε όλε τι πολιτικέ μα προτεραιότητε όπω την ενεργειακή ασφάλεια και τι κλιματικέ αλλαγέ. Την καταπολέμησή του δηλαδή. Από την άλλη, υπάρχουν τέτοιε προτεραιότητε που είναι καθοριστικέ για την ολοκλήρωση τη στρατηγικής ε, του 2020 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάστημα, καινοτομία, έρευνα, τουρισμό. όλα αυτά θα παραμένουν μόνο ωραία λόγια όμως, εάν δεν προβλέψουμε κάτι στο σχέδιο προπολογισμού ήδη για το 2010 λέει Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα. Οι συντονιστές της Επιτροπής ε, Προπολογισμού αποφάσισαν να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια είτε στις 15 ή 16 Ιουνίου. Γι' αυτό πρέπει κατεπηγόντως να ετοιμάσουμε τις τροπολογίες μας και οι δυνατόν με τρόπο ενιαίο. Στη δική μου γνωμοδότηση, στο σχέδιο γνωμοδότησης, προσπαθώ να εντοπίσω ποια είναι τα προγράμματα που ιδιαίτερα ενδιαφέρουν την ΙΤΡΕ και που έχουμε συζητήσει σύντομα στο παρελθόν. Ελπίζω ότι με τι τροπολογίε σας που ήδη έχω συζητήσει με τους Κεώδης και τους πολιτικούς συμβούλους της ομάδας, θα καταλήξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενωμένοι στο να υιοθετηθεί η δική μας συνεισφορά από την Επιτροπή Προπολογισμού. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και η ΤΡΕ και η, η Επιτροπή Προπολογισμού ενώπιον του Επιτρόπου που είναι υπεύθυνο για την έρευνα, την ενέργεια και την ε, βιομηχανίε και να αναλάβουμε πλήρω τα καθήκοντά μα ε, βάσει τι συνθήκε τη Λισαβόνα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα, ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ και τον προσωπικό τη Επιτροπή που ήταν τόσο ευέλικτο να μα δώσουν τη δημοκρατική ευκαιρία να λάβουμε υπόψη ε, τι τροπολογίε και την ψηφοφορία του πριν από την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Προσθέτω επιστρέφονται οι ευχαριστίες σε εσά γιατί κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ο κύριος Μπιουτικόφερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ήθελα Ρίτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε. Με ιδιαίτερο στένος και αλληλέγγυα ως συνάδελφος. Θα ήθελα ταυτόχρονα όμως κάποιες παρατηρήσεις να κάνω για το σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας. και για το ότι ίσως κάποιες ε, αλλαγές μπορεί να υπάρξουν που θα είναι προς μια έκφραση κοινών στοιχείων στην Επιτροπή μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ως πρώτο θα το αναφέρω, αυτό αναφέρεται και στο εδάφιο 3 και είναι η έκρηξη κόστους στο ΙΤΕΡ. Μόλις με τον κύριο Έτιγκερ συζητήσαμε για την έκρηξη του κόστους στο ΙΤΕΡ είναι σίγουρα, δεν είναι τώρα σίγουρα δυνατόν να βρούμε μια δυνατότητα πώς άμεσα θα έχουμε μια, ε, πώς θα αποφύγουμε την κάλυψη του άμεσου κόστους. Όμως ταυτόχρονα και χρηματοοικονομικά δεν θα ήταν λογικό και ευφιές ή και αηφόρο τώρα να ζητάμε νοπό φρέσκο χρήμα και το θέμα του τι θα γίνει σε σχέση με μια περαιτέρω έκρηξη κόστους και την αποφυγή έκρηξης κόστους να μην το καλύψουμε, να το αγνοήσουμε τελείως. Γι' αυτό θα έλεγα τουλάχιστον να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει ένα μηχανισμό που θα λειτουργήσει για τον περιορισμό του κόστους. Όπως, όπως για παράδειγμα στην κοινή αγροτική πολιτική έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό όταν είναι ανεξέλεγκτο το κόστος και οι δαπάνες, ώστε να αποφύγουμε <clears throat> στο πρόγραμμα για την έρευνα για την έρευνα για τα, την ενέργεια να έχουμε μία ας το πω έτσι αμφιβολία για την ε, έρευνα που θα μπορέσει να επιτελεστεί για την έρευνα για την σύνδεξη. Θέλω να υποστηρίξω αυτά τα οποία ανέφερε η συγγήτρια στο σημείο 2 δηλαδή για το ότι μία εύλογη χρηματοδότηση του 7ου προγράμματος πλαίσιου, από αυτή την Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια μ, κατεύθυνση. Και σε σχέση με το σημείο 5 θα ήθελα να προτείνω όταν εκεί γίνεται λόγος για τις υποδομές της ενεργειακές η αναφορά στην αηφόρο ενεργειακή πολιτική είναι ίσως σκόπιμη. Να προσθέσουμε μια τέτοια λοιπόν εκεί αναφορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκας παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας. Συμφωνώ με τις ε, ιδέες που εκφράζονται στην έκθεση Θεωρώ ότι ε, η εργασία που έχει γίνει είναι τεράστια, ε, πόσο μάλλον που το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα κρίσιμο θα έλεγα. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή, ως μέλος του ΕΛΚ, θα έλεγα ότι ε, υπογραμμίζει και τονίζει κάποιες σημαντικότατες προτεραιότητες και υποστηρίζω το έγγραφο αυτό το οποίο έχει υποβληθεί. Όπως είπε ο προαλής σας, εκκρεμούν ακόμα κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, γιατί ε, ο προπολογισμό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε αναφέρει και σε άλλες συζητήσεις στο παρελθόν, ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια ζητήματα ιδίω όταν θα έχουμε πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να λάβουμε πιο ισορροπημένες αποφάσεις και όπως είπε και η συγκήτριά μας, έχουμε ένα πολύ φορτωμένο χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τη μελλοντική μας εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οντί, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγητριά μας για την πολύ καλή της εργασία. Επίσης να θέσω την ε, ακόλουθη ιδέα όσον αφορά την διάρθρωση του προπολογισμού, κυρίως όσον αφορά τη μορφή που θα πρέπει να πάρει αυτή η διάρθρωση. Η φυστάμενη διάρθρωση δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εξελιχθεί προκειμένου να καταφέρουμε να καταχωρήσουμε τις α, τρέχουσες δαπάνες όσον αφορά τις επενδύσεις. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει στα πλαίσια του προπολογισμού του κοινοτικού να έχουμε ένα τμήμα το οποίο να φέρεται στις επενδύσεις όπως ακριβώς έχουμε και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς όπως για παράδειγμα στην Γαλλία στη χώρα μου, στο παράγραφο 6 για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε τέτοια μνήμα και να αναφερόμαστε ακριβώ στι επενδύσει που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα στο πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Γκαλιλαίο δεν καταφέρνει να βρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι είναι τραγικό. Για τέτοια λοιπόν σημαντικά προγράμματα πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα, ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο όσον αφορά τι κοινοτικέ επενδύσει. Αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Επίτροπο στι επενδύσει που θα πρέπει να γίνουν από ενεργειακή πλευρά. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει έρθει πλέον η κατάλληλη στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, να έχουμε στον επίσημο κοινοτικό προπολογισμό ένα τμήμα που θα αναφέρεται ξεχωριστά σε επενδύσει. Να αναφέρονται δηλαδή επενδύσει ξεχωριστά από τι τρέχουσε δαπάνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλοι να ζητούν τον λόγο. Θέλετε εσεί και πάλι. Παρακαλώ, Herzog. Ε- πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τι πολύ καλέ συμβουλέ που μου έδωσαν και περιμένω και τι τροπολογίε σα. Θα ήθελα να κάνω μία παρατηρήση σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριο Σοντή. Συμφωνώ με την άποψή σα. Όντω, τα προγράμματα αυτά για την διαστημική έρευνα και τον Desert και τον Ναμπούκο ανοίγουν ένα εντελώ καινούριο κεφάλαιο στι υποδομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για κοινοτικέ πλέον υποδομέ που στείνει και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σα, αλλά θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Αν θα καταφέρουμε να έχουμε και συλλογή τελών αν θα έχουμε εισφορές ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές αυτές υποδομές και πώς θα καταφέρουμε να τις εντάξουμε τις ενδεχόμενες αυτές μελλοντικέ εισφορές στον κοινοτικό προπολογισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ <clears throat> υπενθυμίζω για την προθεσμία 11 Μαου. θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα επόμενο σημείο 9 περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργία θέσεων ε, μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμη οικονομία, αηφόρου οικονομία. Η κυρία Φιγκερέδο, η συγγήτρια, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Έχετε τη σειρά τώρα, κυρία Φιγκερέδο, εσεί. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξεπώνησα, όπως μπορείτε να δείτε, επτά προτάσεις ε, που θεωρώ ότι έχουν τη σημασία τους υπό το πρίσμα της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιομορφίες κάθε κράτους μέλους και του βαθμού της ανάπτυξης των βιομηχανιών κάθε κράτους μέλους και την γνώση που υπάρχει σε σχέση με κάποιους τομείς, καθώς επίσης και τις ανάγκης που υπάρχει να προασπίσουμε την απασχόληση εκεί και το περιβάλλον επίσης. Επίσης μετά να λάβουμε υπόψη ότι οι λύσεις κυρίως στον τομέα της καινοτομίας αλλά επίσης και στον τομέα της καινοτομίας, της βιομηχανικής καινοτομίας πρέπει να δίνουν απαντήσεις να δίνουν απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα τα οποία ζούμε και αντιμετωπίζουμε και που έγιναν ακόμα πιο πιεστικά μέσα σε μια περίοδο κρίσης όπως η ανεργία, η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η υπεργύρανση του πληθυσμού, η σπανίδα των ενεργειακών πόρων και γι' αυτό όχι μόνο υπάρχει ανάγκη να υποστηρίξουμε τη δημόσια έρευνα και το να, διαθέσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στις μικρές, μεσαίες και, μικρο, και πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά εξίσου να λάβουμε υπόψη και την ενεργειακή αποδοτικότητα και απόδοση με νέους, νέες πηγές ενέργειας ως πόρο, αλλά και νέες διαδικασίες παραγωγής, ανακύκλωση, καλύτερη εκμετάλλευση πόρων. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη στόχο, πάντα έχοντας υπόψη ως στόχο, όχι μόνο να διασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε την απασχόληση, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης με αηφορία σε άλλους τομείς, στους ίδιους τομείς ή και σε νέους τομείς, βιομηχανικού τομείς για παράδειγμα, με τρόπο ώστε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε, την ανεργία και την αποβιομηχανοποίηση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις περιφέρειες που είναι θύματα αυτής της αποβιομηχανοποίησης σε κάποιες περιπτώσεις επειδή είχαν μεγάλη συμπίκνωση βιομηχανικών τομέων και πλήγησαν ιδιαίτερα, μια και βρέθηκαν σε κρίση αυτοί οι τομείς. φαντουργία για παράδειγμα ή και για τα αυτοκίνητα, αυτοκινητοβιομηχανία επίσης και σε άλλους τομείς ε, <clears throat> όσον αφορά αυτή την κρίση. Επίσης και αυτοί να ληφθούν υπόψη. Η μετεγκατάσταση πολυεθνικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, κυρίως από την Πορτογαλία στο εξωτερικό που είχε πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις σε πολύ μεγάλες ζώνες στην περιφέρειά μας. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί υποστήριξης και ανακούφισης και υποστήριξη της, της καινοτομίας και της απασχόλησης, ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες ε, και να... οι περιφερειακές ανισότητες. Στον τομέα της αποδοτικότητας, ε, στον τομέα της ενέργειας, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες από την ε, τον οικοδομικό τομέα μέχρι τις βιομηχανίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις απασχόλησης απασχολώντας, αναπτύσσοντας τομείς που είναι θεμελιώδεις. Θεμελιώδης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Κυρίως υπάρχουν χώρες όπου η κατάσταση αυτή είναι πιο πιεστική και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και όπως είχα ευκαιρία να πω <clears throat> σε σχέση με τον Επίτροπο, Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης στον τομέα των ενεργειακών τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν και η ενεργειακή φτώχεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυξάνεται αυτό το πρόβλημα σε διάφορες χώρες μας. Επίσης πιστεύω κατά τα άλλα ότι εδώ μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης με την έρευνα. Με την έρευνα και επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς που θα δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα μετά από τις αλλαγές και μεταβολές που είδαμε στο παραγωγικό τομέα πρέπει να συνοδευτούν με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με την διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Όλα αυτά πρέπει να προγραμματιστούν και να σχεδιαστούν όπως πρέπει να προγραμματιστούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κάθε χώρα και στην περιφέρεια στους δήμους και κοινότητες και στο τοπικό ακριβώς επίπεδο για να μην δημιουργούνται μεγαλύτερες ανισότητες και μεγαλύτερες ασημέτριες και να μην έχουμε μεγαλύτερη απώλεια θέσεων απασχόλησης αντί να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Σε αυτούς τους τομείς, όλους αυτούς τους τομείς, υπογραμμίζω τη σημασία του δημόσιου τομέα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση που θα είναι πιο αηφόρα. Είτε υπό όρους απασχόλησης, είτε υπό <clears throat> καταπολέμησης της φτώχειας, είτε ακόμα υπό τους όρους της καταπολέμησης των ανισοτήτων και των ασυμμετριών, περιφερειακών και τοπικών. Γι' αυτό για όλους αυτούς τους τομείς, ενέργεια, στην δημιουργία υποδομών, εξοπλισμού, μεταφορών, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών, είναι όλοι αυτοί οι τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης. Πρέπει όμως <clears throat> να τις χειριζόμαστε με τις αποτελεσματικές ε, δημόσιες πολιτικές και να τις κατευθύνουμε με τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Αυτές είναι οι προτάσεις μου στη γνωμαδότησή μου και αναμένω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέφων. Ευχαριστώ. Ε, als nächstes Tänan ja olen Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τη συντάκτρια γνωμοδότησης για το έγγραφο αυτό και συμφωνώ με πολλές πτυχές αυτής της γνωμοδότησης. Τούτου λεχθέντος αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και αυτό απαιτεί εκβάθρον σημαντικές αλλαγές στις βιομηχανίες μας. Δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το θέμα της μείωσης ε, της χρήσης πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους πιο αποτελεσματικά, ώστε οι βιομηχανίες μας να ακολουθούν μια πιο ε, αηφόρο πορεία. Επίσης, να προαγάγουμε την καινοτομία. Αυτό σημαίνει ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει δυνατότητες παράλληλων δράσεων, που πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τώρα, <clears throat> βράχει πρόθεσμα. Πού πρέπει να επικεντρωθούμε. Στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Μέσω πρόθεσμα πρέπει να αποφύγουμε να χρησιμοποιούμε υψηλές εκπομπές ρήπων ε, τεχνολογία ή πηγές ενεργειακές και μακροπρόθεσμα να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με την ε, βιομηχανική μας προσπάθεια και να είμαστε προσεκτικοί στην διαχείριση φυσικών πόρων. Τώρα, σήμερα πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε πώς όλες αυτές οι αλλαγές θα πάρουν σάρκα και οστά χειροπιαστά και θα εφαρμοστούν. Οι αλλαγές για τις οποίες κάνω λόγο δεν, είναι, δεν προωθούνται απλά <clears throat> από την ΚΑΠ ή από το, ενεργεια... το πρόγραμμα για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη, το επταετές πρόγραμμα ή άλλα προγράμματα. Είναι ατομικές, εξατομικευμένα μέτρα, αλλά δεν επαρκούν μια και υπάρχει αναγκαία επίγουσα επιτακτική ανάγκη για αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουμε. Με άλλα λόγια, τι σημαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και να αλλάξουμε το υφιστάμενο πλαίσιο. Χρειαζόμαστε καινούρια πλαίσια, όπως τέλη για το περιβάλλον και την οικολογία, εκοτάξες. Επίσης χρειαζόμαστε <clears throat> έρευνα όσον αφορά τις βιομηχανίες μας και τους ερευνητές μας που πρέπει να συνεργαστούν ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκμετάλλευσης αυτών των πόρων. Για παράδειγμα, σε σχέση με κτίρια που πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν αλλαγές ώστε να προσαρμοστούμε με τις, στις ανάγκες. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα είναι σημαντικός ο ρόλος των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σε θέση να ακολουθήσουν αλλαγές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως μπορεί να θεωρούν τον εαυτό τους ασήμαντο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν όλες όμως συνενωθούν και δράσουν από κοινού σε ένα ενιαίο πλαίσιο μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες αλλαγές. Θα καταθέσω τροπολογίες ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Κύριο Ζαντό, επόμενος αγορητής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, το επίπεδο της κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη μας αναγκάζει να βάλουμε και το κριτήριο της απασχόλησης όλο και περισσότερο σε αποφάσεις που κάνουμε για την ενέργεια και τη βιομηχανία. Και ως προς αυτό, η εργασία που έχει κάνει η συγγήτρια πραγματικά κινείται στο σωστό δρόμο. Θα θέλαμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή με κάποια επιπλέον σημεία. Πρώτον, να εγγυηθούμε ότι η βιομηχανική πολιτική θα είναι σαφής και ότι θα ακολουθεί ουσιαστικά τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να καταφέρουμε να έχουμε στις πολιτικές αυτές όλα τα διοικητικά, φορολογικά στοιχεία της πολιτικής που ακολουθείται από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο βιομηχανικό τομέα. Η συγκέντρια επιμένει πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Ωστόσο, Πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλέψουμε άλλους προσανατολισμούς όσον αφορά την παραγωγή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε κάθε κράτος μέλος, να υπάρχει μία υποστήριξη προς την ε, ταυτοποίηση και άλλων ε, τομέων δραστηριότητας. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία είδαμε ότι υπήρχε μια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει από εμάς η κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να εγγυηθούμε τις θέσεις εργασίας. Επίσης βλέπουμε ότι σε μεγάλους τομείς που έχουν ε, πάρα πολλούς εργαζομένους, όπως για παράδειγμα στα δηληστήρια ή στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα πλαίσια των μεγάλων αυτών επιχειρηματικών ομίλων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σοβαρή συζήτηση για τον προσανατολισμό που ακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές τόσο από πλευρά εργοδοσίας όσο και από πλευρά συνδικαλιστικών οργανώσεων δηλαδή πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις αυτές σε 10, 15, 20 χρόνια και πώς ουσιαστικά θα υποστηριχθούν στη διάρκεια αυτή οι ε, εργαζόμενοι. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, αν θέλουμε να εντάξουμε περισσότερο τη διάσταση της απασχόλησης στην πολιτική μας, να καταφέρουμε να δούμε σε κάθε τομέα ποια είναι η ε, ένταση απασχολησιμότητας, αν θέλετε, δηλαδή πώς, ε, ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων και πώς θα εξελιχθεί. Για παράδειγμα, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, επομένως θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν για χάρη της κοινωνικής Ευρώπης να ενσωματώσουμε τα κριτήρια αυτά στην πολιτική μας. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα σκεπτικισμός αυτή τη στιγμή, ιδίω όσον αφορά το κλίμα. Μέσω από μια ισπανική μελέτη είδαμε ότι υπάρχει ένα σκεπτικισμό όσον αφορά την δημιουργία πράσινων θέσεων εργασία. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια τη Επιτροπή μα να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή για να μην χάσουμε και άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν, παρακαλώ. Όχι. Τότε ολοκληρώνουμε α, για σήμερα αυτό το σημείο στη μέση διατάξη. 11 Μαΐου επισημένο, 12 το μεσημέρι, προθεσμία 11 Μαΐου 12 το μεσημέρι προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Η κυρία Σιγήτρια όμως θέλει να πει δύο λόγια. Παρακαλώ, συγγνώμη κυρία Φιγερέδο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ολοκληρώσω. Γενικά συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Και φυσικά ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης για την αποστολή γραπτών προτάσεων τροπολογιών, ώστε έτσι να, βελτιώσω, να υπάρξει βελτίωση της ε, ε, γνωμοδότησης. Ε, όμως, επίσης, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δώσουμε κάθε προσοχή, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε βιομηχανικές πολιτικές που θα είναι σαφείς, θα έχουν διάρκεια και αηφορία. Πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει αυτή η απέτηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως εξίσου πρέπει να απαιτήσουμε αυτές οι πολιτικές να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα προβλήματα και τις ιδιομορφίες των περιφερειών μας, των χωρών μας και κυρίως τις ξεχωριστές καταστάσεις οικονομικές και κοινωνικές στις οποίες βρίσκονται και αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες και οι περιφέρειες. Πράγμα το οποίο θα απαιτεί και θα συνεπάγεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. να το κάνουμε αυτό και να επιμείνουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στο, στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Good. Μάλιστα, πολύ καλά. Ακούσατε όλοι. Είναι σαφή η διαδικασία. Ολοκληρώνεται για σήμερα αυτό το σημείο στη ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο 10. Συζητήσεις και παρουσίαση της νέας στρατηγικής ε, του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2010-2020 από τον κύριο Σέγκερ. Σας καλωσορίζω κύριε Γενικέ Διευθυντά για πολλαπλή φορά. Καλώς ήρθατε. Έχετε αμέσως τον λόγο λοιπόν και οι συνάδελφοι θα σας παρακολουθήσουν με κάθε προσοχή. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Τόσο σύντομα μετά την προηγούμενη παρουσίαση μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη νέα στρατηγική μας συνεργασίας. Θα θυμάστε ενδεχομένω ότι είχαμε ένα πάνελ με τον Sir David King που έκανε κάποιες συστάσεις. Μεταξύ αυτών ότι θα πρέπει να φέρουμε την οργάνωσή μας σε ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσμάτων, να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική και ένα νέο όραμα για τα επόμενα έτη, προκειμένου να διεξάγουμε καλύτερο τρόπο την δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε. Βλέπω και τις διαφάνειες που έχω φέρει μαζί μου. Βλέπετε εδώ πέρα πώς θα διαρθρωθεί η παρουσίασή μου. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση και θα περάσω στην ουσία. Δεν θα ήθελα να καταναλώσω πάρα πολύ χρόνο. Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε από επιστημονικής και τεχνικής πλευράς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κατά νου τον Ευρωπαίο πολίτη και τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν τα καλύτερα κέντρα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο παρελθόν και Ξέρουμε πλέον ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε την αποστολή μας, ενδεχομένως να την τροποποιήσουμε σε τρία χρόνια, όταν δηλαδή θα έχουμε επιτύχει να καλύψουμε όλες τις προκλήσεις εκείνες που έχουμε στο, στην αρχική μας δήλωση, στη δήλωση του οραματός μας δηλαδή, όπου λέγαμε τι θέλουμε να γίνουμε μέσα σε τρία χρόνια και θα έρθω αργότερα στο σημείο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ορίσουμε αυτή τη στιγμή από την αρχή το λόγο ύπαρξή μας και την αποστολή μας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε περίπου 700 επιστήμονες που συνεργάζονται μαζί μας, έχουμε πάνω από 400 φοιτητές σε επίπεδο διδακτορικού, Έχουμε λοιπόν τη συμβολή πολλών νέων ανθρώπων, ανθρώπων που έρχονται σε εμά μέσω των προγραμμάτων κινητικότητα σπουδαστών προκειμένου να μας βοηθήσουν, προκειμένου να συνεργαστούν μαζί μας. Το πιο σημαντικό για μας βέβαια είναι να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις για το ζήτημα αυτό. Το σημαντικό πάντως είναι ότι συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές οργανώσεις παγκοσμίως η χρηματοδότησή μας είναι 85% από τα προγράμματα πλαίσιο, 15% είναι, τα, ισο, έσοδα τα οποία έχουμε, που ήταν πέρυσι 6 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς διαχειριζόμαστε τις υποδομές μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν νοικιάζουμε κτίρια, χτίζουμε και διαχειριζόμαστε εμείς τα κτίρια και τα εργαστήριά μας και τα πυρηνικά ε, εργαστήριά μας και με ιδιαίτερη περηφάνεια λέω ότι είμαστε ενδεχομένως ε, η ε, καλύτερη, αν θέλετε, υπηρεσία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα, ως προς την ποιότητα. Καλύπτουμε πάρα πολλά πιστοποιητικά ISO και έχουμε πολλά εργαστήρια τα οποία έχουν επιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πιο αυστηρά τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιοτικής διαχείρισης. Βλέπετε και στη διαφάνεια, διαφάνεια ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής μας. Βασικός στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις κοινοτικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Αναφέρομαι λοιπόν εδώ πέρα στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη επίση ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούμε με πολύ περισσότερα ζητήματα σε κοινοτικό επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε και την ίδια μας την οργάνωση. Πώς καταφέρνουμε τελικά να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μεμονωμένα αυτή τη στιγμή μόνο στον επιστημονικό, τεχνολογικό τομέα. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολυεπιστημονικοί και να καταφέρουμε να κινηθούμε και σε νέους τομείς, να καταφέρουμε να αποκτήσουμε κάποιες νέες αρμοδιότητες. Αυτό λέγεται και στην έκθεση King, δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο κατά νου τον καταναλωτή, τον πελάτη. Θα πρέπει πολλές φορές να αναλάβουμε προορατική δράση και να καταφέρουμε να ταινίσουμε περισσότερο το μέλλον προκειμένου να προκαταλάβουμε κάποιους κινδύνους, κάποιες προκλήσεις που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Και προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γρήγορα για να προστατεύσουμε τον πολίτη εφόσον αυτό κρυφθεί αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε κάποιες αναλύσεις κόστους-οφέλους στις ε, επιλογές πολιτικής που κάνουμε. Βάσει λοιπόν όλων αυτών των απαιτήσεων, καταλήξαμε σε μία νέα δήλωση οράματος. Ουδέποτε είχαμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν, τώρα όμως το έχουμε. Ήρθαμε σε επαφές με πολλούς από τους πελάτες μας, τους ρωτήσαμε τι θέλουν να δουν από εμά και ουσιαστικά θέλουν να τους δίνουμε κάποιες επιλογές οι οποίες να τεκμηριώνονται επιστημονικά προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον καλύτερες κοινοτικές πολιτικές. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μεμονωμένα κράτη-μέλη, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο και θεωρούν όλοι ότι αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Πώς θα καταφέρει βέβαια το κοινό κέντρο ερευνών να εντοπίσει τις καλύτερες επιλογές πολιτικής. Θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο διάλογο με τις Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την, εξ από την πρώτη φάση δηλαδή κατάρτισης πολιτικής. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει στο παρελθόν και δεν είχαμε καταφέρει να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, είχαμε καταφέρει να εξακριβώσουμε ακριβώς ποιες ήταν οι ανάγκες. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύξουμε μία γκάμα επιλογών πολιτικής και να αναλύσουμε επιστημονικά τα υπέρ και τα κατά. προερχόμενος από ένα καθαρά επιστημονικό περιβάλλον, γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και διάφορες κοινωνικο-οικονομικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει να έχουμε ε, περισσότερες μικρο- και μακροοικονομικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει να αυξήσουμε την, τις δυνατότητές μας, τις ικανότητές μας να κάνουμε ένα καλύτερο modeling για πάρα πολλούς τομείς, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές κτλ. Προσπαθούμε λοιπόν να ταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, να καταφέρουμε να δώσουμε συγκεκριμένε πολιτικέ επιλογέ στους υπεύθυνου χάραξη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορεί να οριστεί τώρα η στρατηγική μα, Υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα που αναφέρονται σε μεγάλεπίβολε στρατηγικέ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από αυτέ. Δεν είναι ποτέ διεξοδικό ο κατάλογο, Αν απευθύνετε σε διαφορετικού αρμοδίου, θα σα δώσουν διαφορετικέ προτεραιότητες. Προσπαθώ στη διαφάνεια αυτή να συμπεριλάβω κάποιε σημαντικέ στρατηγικέ καταρχά η αντιμετώπιση τη Παγκόσμια οικονομική κρίση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, ο ενεργειακό εφοδιασμό κτλ. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε εδώ πέρα και κάποιε άλλε στρατηγικέ. Είμαστε βέβαια ένα οργανισμό με συγκεκριμένου περιορισμού. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα και όλε τι ανάγκε. Ακόμα και οι μεγάλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα κριτήρια και λέμε ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένε προκλήσει, στι προκλήσει αυτέ όπου υπάρχει μια ευρωπαϊκή ή μια παγκόσμια διάσταση. Λέμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με τι στρατηγικέ αυτέ που εντάσσονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και λέμε επίση ότι ε, πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά αν πραγματικά έχουμε τις δεξιότητες και τις αρμοδιότητες για να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο τομέα και αν μπορούμε από ρεαλιστικής πλευράς να ανταποκριθούμε στις αρμοδιότητες που απαιτούνται για τη χάραξη συγκεκριμένη στρατηγικής. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας να αποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές, προσπαθούμε να δούμε στη συνέχεια αν μπορεί να γίνει αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε απευθυνόμαστε σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ας περάσουμε τώρα στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή και ουσιαστικά εδώ πέρα θα αναφερθώ σε αυτό το που ονομάζουμε θεματική χώρη, θεματική τομή του κοινού κέντρου ερευνών. Έχουμε εδώ πέρα δύο συγκεκριμένους τομείς, βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη και ασφάλεια. Βλέπετε στα αριστερά της διαφάνειας ποιοι είναι οι νέοι θεματικοί τομεί με του οποίου ασχολούμεθα. Θέλουμε να κινηθούμε προ μια πιο ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά θέλουμε εδώ πέρα να συγκεντρώσουμε τις οικονομικές ε, δεξιότητες που πρέπει να έχουμε προκειμένου να αποκριθούμε στους συγκεκριμένους οικονομικούς ε, στόχους που έθεσα στην προηγούμενη διαφάνεια. Λέμε επίσης ότι ο, θεματικό, ο δεύτερος θεματικός μας τομέας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τρίτον ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε Μία βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι βασική στρατηγική τομή σε αυτή και έχουμε και εμπειρογνώμονε εξειδικευμένου στου τομεί αυτού. Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο σημαντικό πυλώνα, την ασφάλεια, λέμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με την πυρηνική ασφάλεια, με την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων και την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων και ένα άλλος τομέας που δεν είναι καθαρά στρατηγικός είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή μέτρηση των υλικών αναφοράς και χρησιμοποιούμε εδώ πέρα πάλι την καλύτερη δυνατή επιστημονική υποστήριξη που έχουμε στη θέση μας. Θα δείτε στο έγγραφο που σας έδωσα περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε στον κάθε έναν από αυτών τους θεματικούς τομείς. Δεν θα επιστέλθω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε προφανώ μπορείτε να θέσετε και κάποια ερώτηση σχετικά. Η περισσότερη θεματική ερευνητική τομή εντάσσονται, όπω σα είπα, στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 και στι σχετικέ πρωτοβουλίε. Παρ' όλα αυτά, συμπεριλάβαμε και κάποιε άλλε στρατηγικέ επιλογέ, όπω για παράδειγμα από τη Γενική Διεύθυνση Προστασία των Καταναλωτών ή από την Γενική Διεύθυνση για την ε, Ασφάλεια των ε, Τροφίμων. Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε να αποκριθούμε τώρα στις προκλήσεις για την συγκεκριμένη στρατηγική. Θέλουμε να συνεργαστούμε με διάφορους φορείς άμεσα και ταυτόχρονα. Αυτό είπαμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θέλουμε να εργαστούμε οριζόντια με διάφορες γενικές διευθύνσεις. Αν η πρόκλησή μας είναι οι κλιματικές αλλαγές, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να συνεργαστούμε θα πρέπει να εργαστούμε όχι καταρχάς βέβαια εμείς στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, αλλά να συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνεργαστούμε και με τους ε, εταίρους μας εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα, κάνουμε μία ανάλυση των ε, δυνατοτήτων που έχουμε σε κάποιους τομείς θα πρέπει να αυξήσουμε τις ε, αρμοδιότητές μας, σε άλλους ε, τομείς θα χρειαστεί να μειώσουμε τις αρμοδιότητες αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να ενδυναμώσουμε την ε, συμβολή μας χωρίς να έχουμε ζητήσει απαραίτητα αύξηση της χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τις πλατφόρμες modeling και τη σχετική εργασία που κάνουμε και λέμε ότι θα κάνουμε πλέον πιο προληπτική εργασία. Στα πλαίσια δηλαδή του κοινού κέντρου ερευνών θα καλούμε τους πελάτες μας από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, θα καλούμε και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα εργαστήρια, σε συγκεκριμένα workshop, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τι θα γίνει για παράδειγμα στη συνθετική βιοτεχνολογία, ποιες είναι τελευταίες εξελίξεις στην γενετική. Υπάρχουν ε, νέοι κίνδυνοι που θα πρέπει να εντοπίσουμε εκ των προτέρων σε αρχική φάση δηλαδή, προκειμένου να ξεκινήσει παράλληλα και μια εργασία που θα μας επιτρέψει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για τους μελλοντικού κινδύνους. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε εκ των προτέρων να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε κινδύνους προτού αυτοί εκδηλωθούν. Ζητήσαμε για αυτόν τον λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσουν ένα κάποιο βαθμό ευελιξίας και να μας επιτρέψουν να προσλάβουμε υψηλά ειστάμενους επιστήμονες στους κατάλληλους τομείς και να υπάρχει μια ευελιξία στην όλη διαδικασία προσλήψεων ουσιαστικά στο κοινό κέντρο ερευνών. Και γι' αυτό τον λόγο χρειαζόμαστε και μια διαδικασία διαχείρισης που θα μας εξασφαλίζει ότι θα καταφέρουμε οικονομικά να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους θεματικούς ερευνητικούς τομείς. Κάποια τμήματα τώρα της στρατηγικής όσον αφορά την εσωτερική διάσταση. Θα καταβληθούν ε, πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για το προσωπικό και τις δεξιότητες. Οι ερευνητικοί οργανισμοί τη σήμερον εποχή, αν πραγματικά θέλουν να κινηθούν στα επίπεδα αριστείας, θα πρέπει να εξελίσσονται γρήγορα, γιατί όλοι εξελίσσονται σήμερα γρήγορα. Είναι λοιπόν σημαντικό να επενδύσουμε σε νέο προσωπικό, στις δεξιότητες του προσωπικού, να προσλάβουμε νέους ανθρώπους εκεί που χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες και θα γίνουν εδώ περισσότερες έρευνες. Επίση, ένα άλλο τομέα που πρέπει να μα απασχολήσει, οι υποδομές και οι ε, κτηριακές εγκαταστάσεις. Όπως σας είπα, δεν έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα στο παρελθόν. Πολλά από τα κτίρια που χρησιμοποιούμε είναι ήδη της δεκαετίας του 60. Ξεκινήσαμε ήδη από πέρυσι να επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο επενδύσεων. 60 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύσουμε σε νέα κτίρια και νέα εργαστήρια και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από ένα μήνα μας έδωσε το πράσινο φως για να γίνουν οι σημαντικές αυτές επενδύσεις. Υποδομές όσον αφορά την τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφοριών. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Χρειαζόμαστε υποδομές γρήγορες, ταχύτατες, με ε, σύγχρονα συστήματα, με πολύ ταχεία μετάδοση πληροφοριών. Επίσης, θέλουμε μια ποιοτική διαχείριση. Θέλουμε να είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος θα επιτρέπει στα εξωτερικά πάνελ να μας εξιολογούν και να βλέπουν ουσιαστικά ότι υποστηρίζουμε τις κοινοτικέ πολιτικές. Θέλουμε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή διασφάλιση της ποιότητος. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο ουσιαστικά και για τους πελάτες μας, ότι ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις απαιτήσει τους. Και τέλος έχουμε και ένα σύστημα διαχείρισης της γνώσης. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δεν κάνουν τα δέοντα στον τομέα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δουλεύουν στους οργανισμούς για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά φεύγουν και παίρνουν μαζί τους και την υπερογνωμοσύνη τους. Αρχίσαμε λοιπόν να διεργαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα προκειμένου η γνώση η οποία δημιουργείται στον οργανισμό να μένει στον οργανισμό μας, να μένει στο κοινό κέντρο ερευνών και να, την, να από αυτήν όλοι. Τώρα, περνάμε στην εξωτερική διάσταση. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μια στενή συνεργασία και εταιρική σχέση με σημαντικούς οργανισμούς σε διάφορα κράτη-μέλη. Θα υποστηρίξουμε την διεύρυνση και την ελοκ ολοκλήρωση σε όλη την επικράτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολύ καλή φήμη στις υποψήφιες χώρες και τις βοηθάμε να φτάσουν το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την επιστημονική τους νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας. Βλέπετε εδώ πέρα ένα διεξοδικό κατάλογο πολιτικών που υποστηρίζουμε. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πάλι διάσταση, θα υποστηρίξουμε τις βασικές προτεραιότητες του Επιτρόπου μας όσον αφορά την καινοτομία. Έχουμε δύο Ινστιτούτα, δύο σημαντικές ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στην Task Force του Επιτρόπου μας για να υποστηρίξουμε την ατζέντα καινοτομία και για να βοηθήσουμε την Ευρώπη να εξελιχθεί σε μια καινοτόμα οικονομία. Τέλος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάω ότι βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να μιλήσω και για εσά. Είστε ένας από τους σημαντικούς παράγοντες βλέπετε ότι εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώνουμε, για το τι κάνουμε, για το που κινούμεθα. Σας ενημερώνουμε εγκαίρως για όλες τις δραστηριότητές μας, για το πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας. Ανταποκρινόμαστε επίση στις απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει μελέτε για σας, συμμετέχουμε στη ΣΤΟΑ. Κάθε φορά που μα καλείτε στη ΣΤΟΑ πηγαίνουμε και φέρνουμε μαζί μα και επιστήμονε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή ομάδα εργασίας που υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Interface Working Group, και κατά αυτόν τον τρόπο μέσω της ομάδας αυτής να σας διοχετεύουμε πληροφορίες και μπορείτε εσείς μέσω της ομάδας αυτής να υποβάλλετε αιτήματα και ερωτήματα προς εμάς. Θέλουμε να διατηρήσουμε την συχνότητα αυτή επαφών που έχουμε και επισκέψεων που έχουν κάνει πάρα πολλοί ευρωβουλευτέ ήδη προ τον δικό μα οργανισμό. Το καλύτερο δυνατό πρέπει να κάνουμε, η καλύτερη εγγύηση, αν θέλετε, τη συνεργασία μα είναι η στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλο, πρωτού ολοκληρώσω και πρωτού που βέβαια σε ερωτήσει σα, να σα προσκαλέσω στο εξή. Ξέρετε ότι σήμερα θα εγγενιάσουμε μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6.30 παρουσία του Επιτρόπου και του της Επιτρόπου Γκέγγεν Κίν, με συγχωρείτε, και της α, Αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Διάννα Γουόλης, Όλοι οι διευθυντέ από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και πολύ σημαντικοί επιστήμονε από τον οργανισμό μα θα είναι παρόντε στην έκθεση αυτή. Σα καλώ λοιπόν να έρθετε προκειμένου να συνειδητοποιήσετε τι κάνουμε σε διάφορου τομεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κορέρα Ντεκάμπος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σέγκελ. Είναι μια από τις πολλές φορές που συναντιόμαστε. Ίσως είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που βρισκόμαστε. Και αισθάνομαι ότι υπάρχει πρόοδος στην ανάπτυξη των ιδεών, εάν μπορώ να το πω έτσι. Πιστεύω από την άποψη την ενοιολογική έχουμε κέρδη σε αυτό το βραχή διάστημα των έξι μηνών. Όπου εγώ ως μέλος της ομάδας διαπαθής GRC έχω αναλάβει καθήκοντα και συμμετάσχω στην διαχείριση της ομάδας αυτής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή σας και για τη σαφήνεια με την οποία μας παρουσιάσατε τόσα συμπυκνωμένα στοιχεία με τόσο ουσιαστικό περιεχόμενο. Να τονίσω ότι Έχουμε εδώ μια αλλαγή, μια σαφή αλλαγή θεώρησης. Η πρώτη θεώρηση, η προηγούμενη μάλλον, ήταν βασισμένη στις ανάγκες του πελάτη και περιοριζόταν στις επιστημονικές και τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες κατά τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όμως αυτή τη φορά το αίτημα για μια νέα θεώρηση είναι και μια, ένα αίτημα για νέο πολιτικό προσανατολισμό, ώστε το κοινό κέντρο ερευνών να κινητοποιηθεί για να ορίσουμε πολιτικές ε, πλέον. Βεβαίως, συστάσεις, αναλύσεις, μελέτες ε, εξωτερικών συνεργατών μας έχουν δείξει τα ίδια στοιχεία, όπως εκείνη του, καθηγητά του καθηγητή David King. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν είναι πολύ επικοδομητική, πολύ ενδιαφέρουσα και όπως υπογραμμίσατε οι προσπάθειες να σπάσουμε τον αποκλεισμό κάποιων θεσμικών οργάνων, η προσπάθεια να εντάξουμε και να ενώσουμε τις προσπάθειες των γενικών διευθύνσεων, να ακολουθήσουμε μια οριζόντια προσέγγιση, όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά επίσης, παρόλο που όλα αυτά είναι σημαντικά, υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα, υπάρχουν και κίνδυνοι. Για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές διαβουλεύσεις, Πρέπει να έχουμε μια ευρεία θεώρηση των πραγμάτων. Βεβαίω, η δράση του Κοινού Κέντρου Ερευνών βασίζεται σε 7 τομεί, κεντρικού τομεί των ε, δραστηριοτήτων του. Εδώ, ίσως είναι δύσκολο να εμπλέξουμε αυτούς τους τομείς τους πολιτικούς μας προσανατολισμούς ή να προσαρμόσουμε τους πολιτικούς προσανατολισμούς σε τομείς όπου δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Η μεγαλύτερη δυσκολία που βρίσκω να υπάρχει στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής είναι στην ποσοτική καταμέτρηση των στόχων, των, των συγκεκριμένων στόχων. Μας είπατε ότι θα προγραμματιστούν νέοι στόχοι, υπάρχουν ήδη νέοι στόχοι και χρειάζονται δείκτες πιο συγκεκριμένοι, οι οποίοι να μπορούν να ενταχθούν, να καταμετρηθούν ως προς την ποσότητα και να ενταχθούν σε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια μέθοδος μέτρησης Καινούργια, διαφορετική από αυτή με την οποία αξιολογείται ένα οποιοδήποτε ερευνητικό Ινστιτούτο. Αυτή λοιπόν η μέθοδος μέτρησης θα πρέπει να μελετηθεί. Ωραία θα ήταν να μας κατεφέρει ήδη κάποιους δείκτες αξιολόγησης, αλλά προφανώς υπάρχει εδώ ένα σημαντικό έργο που πρέπει ακόμη να γίνει. Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ υπάρχει μια μικρή αμφισημία, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω αυτή την αδυναμία. Γιατί, κύριε Σέγκελ, λέτε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία στον συντονισμό του προσωπικού. Συμφωνούμε περισσότερο από ποτέ. Όμω, από την άλλη, πρέπει να ξέρουμε ότι το γεγονό ότι 7 θεσμικά όργανα ή το 85% της χρηματοδότηση των θεσμικών αυτών οργάνων προέρχεται από κοινοτικού πόρους, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει υπέρμετρη ηρεμία, υπέρμετρος καθησυχασμός. Δεν υπάρχει αρκετή κινητοποίηση για την έρευνα. Ε, και η ανταγωνιστικότητα εδώ δεν ξεχνάμε ότι είναι καθοριστική σημασία για την εξέλιξη όλων αυτών των στοιχείων. Πώ λοιπόν πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία, να κερδίσουμε ευελιξία, στο συγκεκριμένο πλαίσιο από το οποίο ξεκινάτε, με ερευνητέ που έχουν πια το καθεστώ ε, του μονίμου υπαλλήλου. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν και παχυλούς μισθούς. Η χρηματοδότηση λοιπόν, εδώ περίμενα η νέα ε, αποστολή, η νέα εντολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών ήταν πιο φιλόδοξη λόγω της εξωτερικής χρηματοδότησης. Λέτε ότι το 15% της εξωτερικής χρηματοδότησης παραμένει. Δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό το όριο δεν υπάρχουν ενδείξεις να υπάρχει διάθεση να ξεπεραστεί αυτό το όριο, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια σχετική τελμάτωση, μια παραμονή στο status quo, στην άνετη ζωή στην οποία έχετε συνηθίσει. Πολλά εργαστήρια εξωτερικά ακόμη και κρατικά έχουν πολύ λίγα εξωτερική χρηματοδότηση, ούτε καν 15% τα περισσότερα από αυτά σήμερα ουσιαστικά σκοτώνονται στη δουλειά, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κερδίσουν κάτι. Και για να ολοκληρώσω, ένα μικρό πρόβλημα συνέπειας κατά την άποψή μου. Εντόπισα τους τομείς προτεραιότητάς σας. Είπατε ότι πρώτος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική και μακροοικονομική πολιτική, ε, η εκπαίδευση, η χαμηλή καταναλωσία άνθρακα, η βιώσιμη διαχείριση των ε, πόρων. Και μετά είπατε την ασφάλεια, safety and security. Και βεβαίω μια ενιαία αντιμετώπιση για την πυρηνική ασφάλεια. Όμω, όταν προτείνετε την ε, πρικοδότηση από τον προπολογισμό στο λίμα ασφάλεια επισητιστική από 18% σε 12%. Στην πυρηνική ασφάλεια παραμένει το 22%. Και στο ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων προτείνεται μείωση από το 14% στο 11%. Αυτές οι μειώσεις στον προπολογισμό, αυτές οι περικοπές πιστεύετε ότι συνάδουν με το στόχο σας να ενισχυθεί η ασφάλεια, safety and security να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την διάβγεια της ομιλίας σας, διότι αυτή η θεώρηση είναι πραγματικά καινούρια και χαράζει νέους δρόμους για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Ένσου. Ευχαριστώ τον κύριο Σέγκελ για την παρουσίασή του. Εκτιμούμε την, το έργο του Κοινού Κέντρου Έρευνας, γιατί πραγματικά στηρίζει από τεχνικής και επιστημονικής άποψης και εμάς που πρέπει να το εξεργαστούμε και να σχεδιάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας. Εξ όσων κατάλαβα, το κέντρο σας έχει σημαντική ερευνητική υποδομή. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσατε να έχετε καταλήξει στα τόσο θετικά αποτελέσματα που και εσείς μας περιγράψατε. Και ειδού το ερώτημά μου. Τι πιστεύετε για τις ανάγκες να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές και στα νέα κράτη-μέλη. Οι υποδομές λείπουν από τα κράτη αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που τα νέα κράτη δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα διευθυντικά ταμεία τα κονδύλια μάλλον προέρχονται από τη διαστοτικά ταμεία και προορίζονται για την έρευνα. Τι συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσατε να κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να βοηθηθούν και τα κράτη που θα έπρεπε να βελτιώσουν τι υποδομέ του. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σέγκελ, νομίζω ότι καταλαβαίνετε γαλλικά. Σωστά. Γαλλικά ή αγγλικά. Ωραία λοιπόν, αγγλικά αν προτιμάτε. Λίγα σχόλια για την ομιλία σας. Για τις θεματικούς τομείς όπου θα επικεντρωθεί το κοινό κέντρο ερευνών. Η επικέντρωση είναι ήδη κάτι. Καλά κάνετε και συγκεντρώνεστε σε στόχους αλλά ήδη θέσατε κάποια ερωτήματα στους εαυτούς σας, ε, όπως φάνηκε, όπως γιατί κάνατε τη μια ή την άλλη επιλογή και μετά αναφέρατε κάποιες προκλήσεις. Μια από αυτές είναι η γύρανση του πληθυσμού, η γύρανση της κοινωνίας. Δεν βλέπω τίποτα στους θεματικούς τομείς όμως για αυτό το σημείο. Η μόνη πτυχή όπου η υγεία σχετίζεται με αυτά που αναφέρατε είναι η πιστιστική αναφερατε ειναι η διασταση Όμως για την βιωσιμότητα, την αηφορία των κοινωνιών μας η ηλικία και η γύρανση είναι σημαντικά ζητήματα. Τι κάνετε λοιπόν γι' αυτό. Και ένα σχόλιο για την ανοιχτή και την ανταγωνιστική οικονομία. Το να δηλώνονται οι θεματικές ενότητες, ήδη αυτό είναι θέμα πολιτικής επιλογής προφανώς. Το θεμελιώδες ερώτημα που θέλω να σας κάνω λοιπόν είναι τι πιστεύετε για την οικονομία, ότι θα πρέπει να έχει σκοπό να αυξάνεται ή να δίνει και κάποιο όφελο στους πολίτες, στους ανθρώπους. Υπ' αυτή την έννοια με ενδιαφέρει η να δινει και καποιο οφελο στους πολίτε, στους ανθρώπου. υπ αυτη την εννοια με ενδιαφερει η αποψη σα. Δηλαδή, εάν οι πολιτικέ μα επιλογέ βασίζονται σε επιστημονικά πορίσματα, οι Ευρωπαίοι φύνοντε για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Δεν θα πρέπει να λάβουν κάποια μέρη, Δεν είναι αυτή η οπτική γωνία που αρμόζει περισσότερο από το να περιγράφουμε μια ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονομία ως αυτό Δεν θέλουμε να δίνει κάποια ωφέλη, να είναι ανταγωνιστική από μόνη της για τον, ως αυτό Και ένα γενικότερο ερώτημα. Στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που έχω ζήσει από τότε που πρώτο ήρθα και ιδίω σε μη εκλεγμένου φορεί όπω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπω ότι σαφώ υπάρχει ένα ζήτημα με την πριτανεύουσα σχολή σκέψη, την φιλο... πριτανεύουσα φιλοσοφία στου περισσότερου τομεί. Εάν δεν υπήρχε, ε, αν υπάρχει μάλλον θεσμικό όργανο που δεν θα έπρεπε να ε, επηρεάζεται από αυτή την ενιαία σκέψη, από αυτή τη μία βασική θεώρηση, θα έπρεπε να είναι το δικό σα το κέντρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλέ επιλογέ και όχι μία. Επιλογέ στον πληθυντικό. Από αυτή την έννοια λοιπόν, εσεί τι κάνετε ω πρόεδρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών για να βεβαιωθείτε ότι οι προσλήψει, η διαδικασία προσλήψεων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους, σε εργαζόμενους μάλλον που έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, να εργαστούν σε εσά. Η οικονομία, μια σημαντική πτυχή, είναι κάτι που ξέρουμε ότι πλέον στον 21ο αιώνα ε, οδηγείται σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Καθορίζεται το μοντέλο αυτό από το ότι αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς, ε, που, τα όρια του πλανήτη μας. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στους ε, θεματικούς αστομείς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και την οικονομία και όλε τι πολιτικέ σα επιλογέ με διαφορετικέ φιλοσοφίε από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Είναι λίγα τα ακαδημαϊκά κέντρα, τα πανεπιστήμια που ε, προσφέρουν ερευνητέ που είναι εκπαιδευμένοι να έχουν διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Δεν κατακρίνω το κοινό κέντρο ερευνών για τη φιλοσοφία που ακολουθεί, είναι ότι πρέπει να υπάρχει όμω ποικιλία. Και ένα άλλο τομέα είναι η ενέργεια. Με τι γνώσει σα και την πείρα σα εδώ, προφανώ μιλάω στον κατάλληλο άνθρωπο. Εάν θα έπρεπε να δούμε τις ενεργειακές μας επιλογές στην ενεργειακή μας πολιτική. Ξέρετε ότι η συζήτηση για τα πυρηνικά είναι μια συζήτηση που πολλοί είπαν ότι έγινε με βάση τις ιδεολογικές προτιμήσεις και όχι την πραγματικότητα. Και φαίνεται ότι πραγματικά κανείς δεν ε, γλίτωσε από αυτό, ιδίως όσοι ήταν κατά, αλλά ούτε όσοι ήταν υπέρ. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να βασιζόμαστε σε δεδομένα, σε πραγματικά γεγονότα, τη διαχείριση αποβλήτων, την αηφορία τη ε, παροχή, τι γίνεται με τους εργαζομένους που προσλαμβάνει το κοινό κέντρο ερευνών. Τι γίνεται αν όλοι προέρχονται από, την πυρηνική, από τη βιομηχανία των πυρηνικών λόγου χάρη. Δεν θα υπάρχει εδώ προκατάληψη. Αυτό που θέλουμε είναι ε, πολιτικές οι οποίες να προσανατολίζονται σε διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή, να βοηθήσουμε να ανακάμψει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και την πολιτική. Εάν υπάρχουν λίγες πολιτικές επιλογές, σίγουρα το κάθε κόμμα θα προκρίνει τις δικές του, αλλά τουλάχιστον να φαίνεται ότι και τα δύο κόμματα, άσχετα με τις επιλογές που θα κάνουν τελικά, έχουν βασιστεί στα ίδια δεδομένα, τα ίδια στοιχεία. Αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να θέσω. Euh, ο κύριος Σουντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά που ήρθατε μία ακόμη φορά να μας μιλήσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απτύξουμε πιο στενές σχέσεις τώρα που στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε και πιο ενισχυμένε αρμοδιότητες. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε για άλλη μια φορά πώς οργανώνεται η διοίκηση στα πλαίσια του κοινού κέντρου ερευνών πρόκειται για διακυβερνητική τελικά οργάνωση ή είναι κοινοτική η οργάνωση που έχετε. Πάνω από εσά ποιος υπάρχει ουσιαστικά είναι το Συμβούλιο των Διοικητών με επικεφαλής τον κύριο Αλμπίν, τον καθηγητή Αλμπίν, πώς οργανώνει ουσιαστικά διοίκηση. Καταλάβαμε λίγο την μέθοδο, αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιος υπαρχει ουσιαστικα ειναι το συμβουλιο των διοικητων με επικεφαλης τον κυριο αλμπιν τον καθηγητη αλμπιν πως οργανωνει ουσιαστικα η διοικηση καταλαβαμε λιγο την μεθοδο αλλα θα θελαμε να γνωρίσουμε ποιος εχει ε, τις αρμοδιότητες, την πολιτική αν θέλετε εξουσία ανάμεσα στην Επίτροπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο μάλλον των ε, Διοικητών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μοιράζεται ανάμεσα σε όλα αυτά τα όργανα η εξουσία τώρα για τις προτεραιότητες 2013-2020. Πρέπει να σας πω ότι εμεί θέλουμε να πετύχουμε μια πολιτική συνένεση για το ότι ε, θέλουμε να φέρουμε την έρευνα που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινοτικό περισσότερο επίπεδο, να την κοινοτικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Η Επίτροπο, όταν τη θέσε με το ζήτημα αυτό, είπε ότι θέλει να συζητήσει με τα κράτη-μέλη για να δούνε αν μπορούν να προσαρμόσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα. Ποιο ρόλο θα μπορούσε να λάβει στην περίπτωση αυτή το κοινό κέντρο ερευνών και πώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια έρευνα πιο ευρωπαϊκή. Η κυρία Ριέρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέγκελ, Γενικό Διευθυντή του Κοινού Κέντρου Ερευνών, για την παρουσίαση της νέας στρατηγικής του κέντρου για την περίοδο 2010-2020. Η στρατηγική αυτή μας φαίνεται πολύ καλά διαρθρωμένη, ρεαλιστική. παραμένει πιστή στους ε, παραδοσιακούς στόχους του κέντρου και επιδιώκει με το σωστό τρόπο το, την επίτευξη του έργου που έχει ανατεθεί στο κέντρο ερευνών. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Όπως ε, μια από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας, και το σύστημα τη διαλειτουργικότητα, αλλά εδώ, λαμβάνοντα αφορμή από την παρέμβαση του κυρίου Κάμπο, θέλω να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Δηλαδή, πώ περιμένετε σε επίπεδο θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιηθεί το έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Και μάλιστα να σα ευχαριστήσω και για την οργάνωση τη έκθεση που θα γενιαστεί σήμερα το απόγευμα. Πάντω, κύριε Σέγκελ, πιστεύουμε ότι σε γενικέ γραμμέ το Κοινό Κέντρο Ερευνών δεν είναι αρκετά γνωστό ούτε το έργο, τη δουλειά του. Μιλάμε για μια δουλειά συνήθω άριστη. Αλλά δεν προβάλλεται αρκετά. Ούτε αξιοποιείται από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι απαιτεί να γίνουν ε, περισσότερες προσπάθειες, να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη. Αυτό ήταν περισσότερο παρατήρηση παρά ερώτηση. Ευχαριστούμε για το ερώτημα του κυρίου Λάμπερτ. Θέλω και εγώ να βασιστώ σε αυτό για να θέσω το δικό μου ερώτημα για την ισορροπία. Ο κύριος Λάμπερτ μίλησε για την οικονομία. Εσείς μιλήσατε για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές, για το διοξείδιο του άνθρακα. Λαμβάνετε υπόψη τα σχόλια και τα πορίσματα των επιστημών, ε, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει αντίκτυπος, υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με τα διάφορα θέματα που έχετε θέσει στόχου, αλλά δεν συμφωνούν με μία συγκεκριμένη προσέγγιση. Λίγο πολύ, την ίδια ερώτηση με τον κύριο Λάμπερτ είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλού τομεί. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον να σας ευχαριστήσω για όλα σας τα θετικά λόγια και τη στήριξή σας. Το εκτιμώ ιδιαίτερος και βεβαίως το ίδιο και το προσωπικό του κέντρο που παρίσταται. Με μεγάλη τους χαρά θα τα ακούσουν όλα αυτά. Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα ή σχόλια που έγιναν ο κύριος Περίραντε Κάμπος ανέφερε τους δείκτες. Δείκτες που θα επέτρεπαν να, να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις του κέντρου μας. Τρόπον την, τα επιστημονικά αποτελέσματα μπορούμε ούτως ή άλλως να τα αποτιμήσουμε. Διότι υπάρχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπάρχουν πορίσματα αλλά αυτά είναι απλώς δείκτες, είναι ενδείξεις. Δεν μπορεί η επιστημονική πρόοδος να καταμετρηθεί ποσοτικά. Μπορεί όλα αυτά να βοηθήσουν για να κρίνουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα, και αυτό είναι μια πρόκληση, ζήτησα από το προσωπικό να βοηθήσει εδώ, είναι να μετρήσουμε την ε, επίδραση που έχουμε στην πολιτική. Διότι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένω είναι πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την ποιότητα και την, να καταμετρήσουμε όλη την ποιότητα και την ποσότητα της προσφοράς που δίνουμε στους πολιτικούς. Ε, θα έχετε παρατηρήσει πόσα νομικά έγγραφα έχουμε ετοιμάσει, πόσα τεχνικά παραρτήματα, πόσο συχνά γίνονται παραθέματα από τις έρευνές μας. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα γνωστό στον πολιτικό κόσμο. Θα θέλαμε λοιπόν πανευρωπαϊκός να υπάρχει μία μέθοδος ανείχνευσης ε, λόγω χάρη των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Πώς θα καταμετρηθεί αυτό αν έχει επιτευχθεί. Είναι τεράστιο το έργο για να μπορέσουν όλα τα εργαστήρια να συντονιστούν. Όλη η Ευρώπη μαζί να αρχίσει να συζητάει για το θέμα αυτό, να συμφωνήσει μετά στη μέθοδο που να είναι και έγκυρη, να δοκιμαστεί και επιπλέον να βεβαιωθούμε ότι σωστά παρέχεται. Αυτό ισχύει για πολλού τομεί και δεν έχουμε βρει ακόμη τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να καταμετρήσουμε τέτοιου είδου προσφορά. Θέλουμε να το κάνουμε, αλλά θα ακολουθήσω τη συμβολή σα. Θα συνεχίσουμε το ψάξιμο προ στιγμή. Για την ώρα δεν έχουμε καταλήξει κάπου σε κάποια πιστική λύση. Για την ευελιξία. Ελπίζω ότι δεν με παρανοήσατε. Ίσως εγώ εκφράστηκα κακώς. Αυτό που επιδιώκω δεν είναι αρνητική ευελιξία για την ε, προσλήψεις μας. Αυτό που θέλω είναι η Επιτροπή να μας δίνει τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε άτομα με τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για να φέρουν πέρα στους στόχους μας. Η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα από την προδιατίας. Έχουμε ήδη συμφωνία από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την ΕΠΣΟ, την, τον οργανισμό που αναλαμβάνει τις προσλήψεις, ότι θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες προσλήψεις με ε, βασικό κριτήριο τις επιστημονικές γνώσεις, όχι τις γνώσεις management. Θα έχουμε ανεχτούς διαγωνισμούς λοιπόν, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ε, προσληφθούν ως υπάλληλοι, αλλά για συγκεκριμένους τομείς ε, την το σχεδιασμό μοντέλων, την οικονομική πολιτική και ανάπτυξη. Συγκεκριμένε λοιπόν ανάγκε σε συγκεκριμένου τομεί προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο μα. Δεν θέλουμε λοιπόν αρνητική ευελιξία. Μία διαδικασία που να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαίτερε ανάγκε μα και να μα επιτρέψει να διορίζουμε του ταλαντούχου ανθρώπου που θέλουμε. Για το 15% αναφέρατε το 15% επί του εισοδήματο. Δεν θέλω να αντιδράσω υπερβολικά, αλλά όταν το είχα παρουσιάσει αυτό πενταετία ή τετραετία ω ε, μέρος του προγράμματο πλαισίου 7 είχε ζητηθεί και ένα 30% από κάποιου από κάποια κρατημέλη. Εγώ είχα πει κανένα πρόβλημα, αλλά ελάχιστα τότε την εντολή μα. Μην μα ζητάτε να δίνουμε ανεξάρτητη στήριξη στην χάραξη πολιτική και ταυτόχρονα να μα ζητάτε να κερδίσουμε και χρήματα στην αγορά. Διότι η χημική βιομηχανία, εάν το είχα πει αυτό, αν είχα πει ότι για την νομοθεσία REACH θα κάνουμε ό,τι συνεισφορά θέλετε. Δίνουμε τους αριθμούς για οποιοδήποτε ζήτημα σας ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να κερδίσω και λίγα χρήματα. Δεν μπορείτε να μου δώσετε μια ερευνητική σύμβαση για ένα δις. Θα είχα καλύψει το 30% του προπολογισμού μου. Το ίδιο και για, την, για τα τοξικολογικά θέματα, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Εδώ δεν ε, υπάρχει άλλος φορέας που να στηρίζεται πολιτικό στα κάτι μέλη και να είναι σε άμεση επαφή με Υπουργεία και να πρέπει να κερδίσει χρήματα στην αγορά. Άρα λοιπόν με μου τη φέρνετε από την ε, πίσω πόρτα. Δεν ζητάω το κέντρο ερευνών να έχει περισσότερους πόρους, να πρικοδοτηθεί με περισσότερα. Όχι. Καλά λειτουργεί και είναι και ένα σημείο αναφοράς οι υπηρεσίε που προσφέρουμε σε τομεί που στηρίζονται στι αρμοδιότητέ μα και που δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων είναι καθοριστική. Όμω εγώ ε, υπερασπιζόμουν και ο Επίτροπο και ήταν μαζί μου τότε εναντίον κάποιων κατώμελων ήταν το εξή. Δεν μπορεί να γίνουν και τα δύο. Δεν μπορεί να υπάρχει στήριξη τη πολιτική, αλλά να διατηρήσουμε και την ανεξαρτησία μα και ταυτόχρονα να μα ζητάτε να κερδίσουμε και χρήματα στι αγορέ, ή τουλάχιστον πολλά χρήματα, τότε θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Οπότε ε, Παρακαλώ να καταλάβετε καλά το επιχείρημά μου, να καταλάβετε γιατί καταρχήν αποδεχτήκαμε το 15% ως ένα λογικό περιθώριο δεδομένων των ειδικών μας αναγκών και της ειδικής μας αποστολής. Για τον κύριο Ένσου, οι υποδομές στα νέα κρατημέλη δεν μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε από το δικό μας προπολογισμό. Ακόμα και αν το θέλαμε, δεν μπορούμε δεν είναι μέρος της αποστολής μας. Όμως αυτό που έχουμε κάνει ήδη είναι ότι έχουμε προσφέρει στήριξη στα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη και τις χώρες της διεύρυνσης και έχουμε επισύρει την προσοχή των συναδέλφων μας χρόνο το χρόνο μετα, μέσω των διορθωτικών ταμείων ώστε να υπάρξουν επενδύσεις. Επίσης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας να εντοπίσουν το τεράστιο έργο που πρέπει να γίνει ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητε υποδομές στα υποψήφια κράτη-μέλη και τα νέα. Ήδη αρχίσαμε να δορίζουμε εξοπλισμό. Πήγα σε ένα πανεπιστήμιο στη Ρουμανία πριν από πολλά χρόνια και όταν είδα τον εξοπλισμό που διέθεταν, είπα, όταν εγώ έκανα τη διπλωματική μου, πριν από 40 χρόνια περίπου, είχα καλύτερο ηλεκτρονικό, εξοπλισμό από αυτό που έχετε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει γι' αυτό και συμφωνώ 100% μαζί σα. Μπορούμε όμω να στηρίξουμε άλλου συναδέλφου τη Επιτροπή για να το κάνουμε αυτό. Κύριε Λάμπερτ, έχετε δίκιο. Η γύρανση τη κοινωνία είναι κάτι που μα απασχολεί. Δεν έχουμε αποφασίσει όμω να εργαστούμε από αυτού. Είναι προτεραιότητα, είναι πρόκληση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο λόγο είναι ότι απλώ δεν έχουμε αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Όπω τα έχετε δει, έχουμε παράξει στον τομέα της υγείας πολύ λίγα πράγματα, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι δεν είναι σημαντικές εκεί οι αρμοδιότητές μας. Υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες στα κράτη-μέλη και αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν θέλουμε λοιπόν να αναλάβουμε νέες δραστηριότητες, διότι αν δεν είναι σαφής η εντολή, πιστεύουμε ότι άλλοι μπορούν να φέρουν εις καλύτερα το ίδιο έργο. Τώρα, η παρατήρησή σας για την ανοιχτή οικονομία αισθανθήκαμε ότι αυτό ήταν ένα κατάλληλο τίτλο από τη δική μα πλευρά για να στηρίξουμε την ημερήσια διάταξη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη το 2020. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα αναζητήσουμε και δεν θα ερευνήσουμε και τι κοινωνικέ πτυχέ ή τι περιβαλλοντικέ, καθώ και τα άλλα δυνατά τη ημερήσια διάταξη του καταλόγου προτεραιοτήτων. Καταλάβετε το εξή. Δεν σχεδιάζουμε εμεί την πολιτική. Δεν λαμβάνουμε εμεί τι αποφάσει. Και το λέω και στο προσωπικό μα. Ουδέποτε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό με φέρνει και στην άλλη παρατηρήσή σα. Ότι οι επιστήμονε είναι και αυτοί άνθρωποι. Έχουν και αυτοί απόψει. Βεβαίω έχουν και προκαταλήψει. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι κατά πρώτον έχουμε ένα κώδικα συμπεριφορά που ισχύει για τον οργανισμό μα. Κώδικα συμπεριφορά που επιβάλλει κατά την διεξαγωγή του έργου μα να βεβαιωνόμαστε δύο φορέ ότι δεν έχουμε προσωπικά κίνητρα πεπιθήσει ή απόψει που να μα επηρεάζουν. Προσπαθούμε να διασφαλίζουμε την ποιότητα ε, μέσω μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγηση, peer review, ώστε να εξετάζουμε προσεκτικά τα αντικειμενικά δεδομένα. Κάναμε μια έρευνα για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, λόγου χάρη. Εκεί είδαμε από ε, εσωτερική άποψη τι διάφορε πτυχέ. Είδαμε τα επιστημονικά δεδομένα που είχαν ήδη δημοσιευτεί. Είδαμε την, ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ, ποια είναι τα αποδεκτικά στοιχεία ε, γιατί κάποιοι προβάλλουν επιχειρήματα κατά και βάσει ποιών στοιχείων ε, και ποια είναι η ουσία πίσω από όλα αυτά. Πολύ προσεκτικά λοιπόν εξετάζουμε το φάσμα όλων των απόψεων, ακόμα και των επιστημονικών. Διότι κάποιε φορέ τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πολύ λίγα και η αβεβαιότητα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε όσο δυνατόν πιο δίκαιοι και αντικειμενικοί. Όσο γίνεται. Δεν είναι πάντοτε δυνατό αυτό, αλλά δεν είναι και λόγο να σα πω ότι δεν το κάνει κάτι τέτοιο εγώ, διευθυντή τη της, ε, του κέντρου. Όπως είπατε και εγώ τις δικές μου αρμοδιότητες, έχω τις δικές μου γνώσεις και εμπειρίες. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τόσο περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη στο κέντρο μας ώστε να έχουμε την πιο εύρωστη επιστημονική γνώση για την χάραξη πολιτικών. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πόσο εύρωστο είναι το έργο μας λοιπόν. Κύριε Οντή για τις κυβερνήσεις πολύ σύντομα να πω ότι είμαστε ε, διάβλος, απευθείας διάβλος της Επιτροπής. Άρα η γραμμή εντολών είναι πολύ σαφής. Όμως υπάρχει και το Διοικητικό Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη που όμως έχει συμβουλευτικό ρόλο. Δημιουργήθηκε από απόφαση της Επιτροπής. Κάτι σαν προ 15 ετίας. Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Board of Governance είναι να δίνει το πράσινο φως σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που μπορεί να επηρεάζουν την ε, λειτουργία του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Εμπλέκονται τον ε, διορισμό όλων των υψηλών στελεχών. Όχι κανένα μάλλον, κανένας, ε, κανένας διευθυντής δεν μπορεί να διοριστεί πριν να εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό και να λάβει και θετική αξιολόγηση. Είναι λοιπόν συμβουλευτικό το σώμα, αλλά το χρειαζόμαστε στη διαδικασία της Επιτροπής. Νομίζω από όσα γνωρίζω το πολύ δύο ή τρεις άλλοι τέτοιοι διάβλοι έχουν παρόμοια σώματα να το συμβουλεύουν. Τώρα πώς μπορούμε να δώσουμε τη συνεισφορά μας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα πάω στη Σεβίλη με την Επίτροπο για Κουίν αύριο και εκεί θα συναντηθώ ενισχυθούν τα συμβούλια του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ε, συμβουλευτικά ως προς την Επιτροπή και αυτά. Πρώτη προτεραιότητα στην εμμυρίσια διαταξή μας είναι τι μπορεί να κάνουμε, πώς θα συνεισφέρει ε, το Κοινό Κέντρο Ερευνών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Και θα κάνουμε μια γρήγορη επεξεργασία των πρώτων ιδεών, ώστε να δούμε τι μπορούμε να αναπτύξουμε προς όφελος της πολιτική τη Επιτροπή. Έχουν ήδη γίνει πολλέ φιλόδοξε πολιτικέ προτάσει για το πώ θα έχουμε ένα μια καλύτερη ευρωπαϊκή διάσταση και περισσότερη κρίσιμη μάζα προκειμένου να αναπτύξουμε ε, ηγετικού ε, φορεί έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό για να ανταγωνιστούμε τι ΗΠΑ και άλλε χώρε που μα προλαβαίνουν ήδη. Κυρία Μαντουρέλ, το ερώτημά σας αφορούσε τις γνώσεις και την προβολή μας. Το γνωρίζουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι μας γνωρίζει καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον. Πάντως, στα κράτη-μέλη κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσοι μας γνωρίζουν είναι αυτοί που δουλεύουν στα Υπουργεία Έρευνας. Όμως, στην πραγματικότητα, όσοι ωφελούνται περισσότερο από το έργο μας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα Υπουργεία Γεωργίας, τα αντίστοιχα δηλαδή, των γενικών διευθύνσεων που και εμείς ε, εξυπηρετούμε. Δεν εργαζόμαστε για την Γενική Διεύθυνση Έρευνα, ούτε καν για την Επίτροπο που είναι υπεύθυνη για μα. Η συνεισφορά μα τι περισσότερε φορέ είναι επιστημονική τεχνική συμβολή στι χρηματοδοτήσει ε, των διαφόρων πελατών μα, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, τη Γενική Διεύθυνση ε, για την ε, βιομηχανία και ούτω καθεξής. Αυτά δεν είναι πάντοτε γνωστά στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να γίνουμε ορατοί. Αλλά δεν είναι ότι σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχουν και άλλοι φορείς ε, πολύ γνωστοί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Για το δικό σας ερώτημα νομίζω ότι τρόπον την έχω εμέσως απαντήσει. Πραγματικά εξετάζουμε τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν και για τις κλιματικές αλλαγές, Εάν ε, η γεωδυναμική η μηχανική συζητηθεί και αυτά τα συζητάμε, αναλόγω με τι νέε ιδέε που ακούγονται και υποβάλλονται, προσπαθούμε να βρούμε την ουσία στο κάθε θέμα και να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εξέλιξη. Προσπαθούμε να προλάβουμε. Να προλάβουμε τι νέε έρευνε που πρόκειται να ετοιμαστούν παγκοσμίω. Ευχαριστώ. σχόλιο τον κύριο Κατάλαβα την απάντηση που δώσατε στα περισσότερα ερωτήματά μου, αλλά πώς εξασφαλίζεται ότι προσλαμβάνετε εργαζόμενους από πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Έχετε για παράδειγμα πάρα πολλούς οικονομολόγους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί περισσότερο στην νεοκλασική σχολή οικονομίας. Υπάρχουν όμως και οικονομολόγοι που θα μπορούσαν να ακολουθούν Άλλε σχολές. Πώς καταφέρνετε εσεί με του επιστήμονε στους οποίου προσλαμβάνετε να έχετε πολλές οπτικές γωνίε στα πλαίσια του κοινού κέντρου ερευνών. I mean, what, what we do is we watch for scientific... Αυτό το οποίο μας αφορά περισσότερο είναι η επιστημονική ποιότητα και εμπειρία. Δεν συμμετέχω εγώ προσωπικά στις συνεντεύξεις που κάνουμε για τους οικονομολόγους γιατί δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα. Δεν είμαι η στα ζητήματα οικονομίας. Προσπαθούμε πάντως να έχουμε μία εξεταστική επιτροπή η οποία θα εξετάσει την εμπειρία και την ποιότητα την επιστημονική των υποψηφίων. και αν δεν μπορούμε να μετακινήσουμε εσωτερικά εργαζόμενό μας εφόσον δεν έχει την αρμοδιότητα για να μετακινηθεί από τον έναν ερευνητικό τομέα, τον, ε, τομέα στον άλλον, καταφέρουμε πάντα σε εξαιρετικές προσλήψεις. Το βασικό κριτήριο είναι πάντα η αποδεδειγμένη επιστημονική αριστεία στο συγκεκριμένο τομέα. Ζητάμε από τον υποψήφιο να έχει τις δεξιότητες που ανταποκρίνουν ουσιαστικά και στην προκήρυξη της θέσης. Αυτό μπορώ να σας πω. Ελπίζω αυτό να καλύπτει την ε, ερώτησή σας, να καλύπτει την ερώτηση. Να είναι μια πλήρης απάντηση. Πρόεδρος, σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν. Σας καλώ και πάλι αγαπητοί συναδελφοί να έρθετε στα εγγένεια της έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Έκθεση βέβαια η οποία θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επόμενες ημέρες. Η ημερομηνία της διεξαγωγής προσου... της επόμενης συνεδρίασης θα στις 11 Μαΐου. Θα συνεδριάσουμε αρκετά νωρίτερα στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσουμε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες πρέπει να διεξαχθούν εκείνη την